Um, I waiting, hoping we more shadows on Καλησπέρα. Περιμέναμε, περιμένουμε κι άλλο τους σκιώδεις για um, την uh, σκιώδη τραπεζική. Έχουμε όμως uh, τους σκιώδεις της σκιώδους. Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη δεν βλέπω. Ωραία. Άρα εγκρίνεται φαντάζομαι. Έχω πολλές ανακοινώσεις της προεδρου Τρίτη 3η 9 Οκτωβρίου. Υπάρχει αλλαγή στην αίθουσα συνεδριάσεως. Πρέπει να αρχίσουμε στην ώρα μας. Οπότε, αύριο το πρωί συνεδριάζουμε στο PHS 3C50. Αύριο το πρωί. Όχι εδώ λοιπόν, στο PHS 3C50. Αλλά θα επιστρέψουμε αύριο το απόγευμα εδώ, στην σημερινή μας ε, αίθουσα. Η Δίκαιση μας το ζήτησε αυτό. Ε, επειδή κάποια άλλη επιτροπή που είναι έτσι ψηλά ιστάμενη χρειάζεται αυτή τη μεγάλη αίθουσα. Πριν λοιπόν την ακρόαση με τον Μάριο Ντράγκη που αρχίζει στις 9.30 αύριο, στις 9 αύριο το πρωί έχουμε τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με εισηγητή τον Φιλίπ Τεμπάκερ. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων, να είναι αύριο στην αίθουσα που σας είπα στις 9, αλλιώς δεν θα μπορέσουν. Μετά θα έχουμε τη δημόσια κρόαση για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των δημοσιονομικών. Τετάρτη πρωί, 9 με 1, η Επιτροπή θα έχει ακρόαση για αυτό το θέμα. Και οργανώνεται, οργανώθηκε τώρα πρόσφατα όλες οι άλλες αίθουσες είχαν καταληφθεί, οπότε στην 3G2 θα συνεδριάσουμε. Σήτησαμε μεγαλύτερη, αλλά δεν βρήκαμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες στην ASP ε, 3G3, οπότε όσοι προλάβουν θα καθίσουν, οι υπόλοιποι μπορούν μέσω του διαδικτύου να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση για το τριμερή διάλογο και τις οργανισμούς ε, αξιολόγησης πισολυπτική ικανότητας. Τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε με την μόνιμη αντιπροσωπεία για τον πρέσβη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουμε για τους τριμερείς διαλόγους οι οποίοι δεν προχωρούν ικανοποιητικά επί του παρόντος για το CRD4, την οδηγία δηλαδή για την κεφαλαϊκή επάρκεια. Την Τετάρτη που μας πέρασε ήρθε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Οι προσπαθούν να βρουν λύσεις στις διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη του μηνός. Κάποια πρόοδος επιτέθηκε βέβαια στο θέμα της ε, κεφαλαιακής ε, κάλυψης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά πρέπει να υπάρξει κι άλλη πρόοδος αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο να καταλήξουμε μέχρι τα τέλη του μήνα. Επόμενος πολιτικός διάλογος είναι την Πέμπτη και διάφορες τεχνικές ε, συνεδριάσεις έχουν επίσης προβλεφθεί. Για το κάτω, τον τριμερή διάλογο, για αυτό το θέμα συζητιούνται διάφοροι στόχοι και επίπεδα εναρμόνισης στο πεδίο εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι επιλογές των χωρών ομιλών και κάποιες ε, υποχρεώσεις απέναντι στους καταναλωτές. Προχωρούμε πολύ αργά εδώ, ιδιαίτερα στο θέμα του πεδίου εφαρμογής. Η θέση των συνομοδοτών ε, διαφέρουν μεταξύ τους. Και εδώ χρειάζονται τριμερείς διάλογοι. Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί ο χρόνος όσο γίνεται καλύτερα και στον πολιτικό διάλογο για να βρεθούν τεχνικές λύσεις και να συγκλίνουν οι σήμερα αποκλίνουσες απόψεις. 17 και 22 Οκτωβρίου υπάρχουν ημερομηνίες για συνάντηση. Μίλησα πριν για τεχνικό ε, διάλογο. Λάθος έκανα. Τεχνικές ομάδες εργασίες ήθελα να πω. Τώρα τέσσερις ε, συναντήσεις τριμερούς διαλόγου υπάρχουν. Έκθεση κάλετη, ενίσχυση της οικονομικής δημοσιονομικής εποπτείας των χωρών ε, μελών και λιγότερο έχουμε προχωρήσει στην έκθεση Φερέιρα. Τα θέματα που συζητούνται στην έκθεση Φερέιρα είναι πολύ σημαντικά και έγινε, επιτέχθηκε μεγαλύτερη πρόοδο στο τελευταίο τριμερή διάλογο που επικεντρώθηκε στην έκθεση Φερέιρα. Ακούγεται ότι το δίπτυχο πακέτο μπορεί να γίνει τρίπτυχο τελικά. Η Προεδρία και το Συμβούλιο όμως μας είπαν ότι δεν έχουν από το τριμερή διάλογο τέτοια εντολή. Επίσης, επιμένουμε ότι η ποιότητα της τελικής απόφασης ε, πρέπει να διατηρηθεί. Τίποτα άλλο. Πάμε στις σκιώδες, στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Ο εισηγητής έχει το λόγο, Σέιντελ Καντραουή. Παρακαλώ, για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεσή μου έχει 36 τροπολογίες. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για όλες αυτές τις τροπολογίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι προτάσεις τους ήταν κυρίως επικοδομητικές. Εμπληρώνουν το κείμενο, το ενισχύουν, κάτι το οποίο βρίσκω πολύ θετικό. Στόχος μας είναι με τους σκιώδες εισηγητούς να καθίσουμε μαζί και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες, ώστε να διευκολυνθεί η ψηφοφορία που θα γίνει στο Στρασβούργο. Ελπίζω να εγκριθεί τελικά η έκθεση αυτή, οπότε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπως ξέρετε έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, ποιος είναι ο πυρήνας της έκθεσης αυτής. Αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ε, προτάσεις για τον ελεγχό του, πώς εντοπίζονται ε, κίνδυνοι συστημικοί που ελοχεύουν, ποιες είναι οι οντότητες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνει για να ρυθμίσει αυτό το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Νομίζω ότι, εντάξει δεν έχει νόημα όλες τις τροπολογίες να τις σχολιάσω τώρα, αλλά θα αναφερθώ σε κάποιες τουλάχιστον. Διάφοροι συνάδελφοι, για παράδειγμα, ε, αναφέρονται σε ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν κάποιες, δηλαδή ρυθμίσεις υπάρχουν στο σκιώδες αυτό το τραπεζικό σύστημα, αλλά βέβαια άλλες δεν υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν. Και πάνω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη συνάδελφο Βόρτμαν Κόλ, για παράδειγμα 25, που μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για συμβιβασμό. Πάντω οι περισσότεροι συνάδελφοι θα έλεγα ότι ασχολούνται πιο πολύ με το θέμα του ορισμού του Συμβουλίου ε, Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Συμφωνούν οι περισσότεροι ότι πέρα από τη σκιώδη πτυχή του σκιώδους τραπεζικού συστήματος υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Υπάρχουν και θετικέ πλευρέ. Η απαγόρευση του σχεώδου τραπεζικού συστήματο, όπω προτείνει ο συνάδελφο Φέρμπερ, ίσω να μην είναι ότι καλύτερο. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Επίση, χαίρομαι που οι συνάδελφοι Γκουλάρτ, Μπόλ, Κλίν και Λάγκεν στηρίζουν ε, την πρόταση για μια τράπεζα δεδομένων όσον αφορά στοιχεία από το σύστημα αυτό που να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις συναλλαγές ευρώ έτσι ενισχύεται η διαφάνεια. Όπως ε, επίσης μιλούν και για μία ενότητα που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε που να ε, εξετάζει τις ε, μεταφορές οι οποίες ελοχεύουν κάποιο κίνδυνο και αυτό να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Πάλι για την κυρία Βαρτμανκόλ και την κυρία Γκουλάρ θέλω να πω ότι, ναι, συμφωνώ που λένε ότι πρέπει επίση ώρες να είναι το σχεδόν τραπεζικό σύστημα και το κλασικό και να αποφεύγεται το αρμπιτράζ. ότι πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία των συναλλαγών. Το... Ναι, συμφωνώ με αυτό, πρέπει να δουλέψουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Τώρα υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που μιλούν για την ε, οδηγία ε, ανακεφαλαίωσης ε, των τραπεζών, την CRD4 και θέλουν να προσθεθεί και αυτό. Γιατί βλέπουν την οδηγία αυτή, CRD4, σαν ένα πλαίσιο. Τη δυνατότητα να καλύπτει και τις μη τραπεζικές οντότητες Επίσης, στο θέμα της τιτλοποίησης, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή της κυρίας Βάρτμεν Κόλλο και Μπόλς και Κλίνγκς. Να γίνεται τυπλοποίηση. ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις δικές μου τις προτάσεις. Και τέλος, όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια, εδώ συμφωνώ ότι η Ευρώπη δεν είναι μια νησίδα. Πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Γι' αυτό ο κ. Γκάρνερ την προηγούμενη εβδομάδα για τα αμοιβαία κεφάλαια είπε ότι θα υπάρξουν τον Νοέμβριο μεταρρυθμίσεις. Το λέω και εγώ στην έκθεσή μου. Έχει νόημα αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι επίσης θέλουν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια να λάβουν υπόψη τους το USIT 6 που θα ξεκινήσει του χρόνου. Νομίζω ότι μπορούμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν και τα index ε, funds που αποτελούν έναν αδύναμο κρίκο βέβαια. Σύμφωνα πάντως με τις προτάσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Με δύο λόγια. Η αίσθησή μου είναι ότι συμφωνούμε με την γραμμή προς την οποία κατευθυνόμαστε και ότι θα μπορέσουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα να τα συμπεριλάβουμε σε συμβαστικές προτάσεις που θα ετοιμάσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Επικοδομητικά, συνομιλώντας μαζί, ο καθένας θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του και θα καταφέρουμε τελικά να προτείνουμε ένα καλό πακέτο. Ευχαριστώ. Ωραία σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστώ και τον Σάιτ για την εισαγωγή που έκανε σε σχέση με την ε, κατεύθυνση που προτείνει σε σχέση με τις τροπολογίες. Έχω την εντύπωση ότι σε πολλούς κέριους τομείς βλέπουμε να υπάρχει μια σύγκληση ακολουθώντας τη γραμμή που χαράξατε εμείς στην εισαγωγή σας. Για μένα είναι πράγματι πολύ σημαντικό να διακριβώσουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και να μην δούμε μονάχα τους κινδύνους, αλλά να βρούμε και τρόπους καλύτερης ρύθμισης και αποφυγής του να υπάρχει κατάχρηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος για να παρακάμψει κανείς και να αποφύγει τις, ε, ε το ρυθμιστικό άχθος ή την πίεση που μπορεί να προκύψει από την CRD4, την ανακεφαλουργική κεφαλουργικής επάρκειας δηλαδή, ή άλλες ρυθμίσεις. Χρειάζεται λοιπόν το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για να αποτρέψουμε μια τέτοια κίνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν θέλουμε να έχουμε επι, αλληλοεπικαλύψεις ή αντιφάσεις στη ρύθμισή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόταση του κ. Αλχάντραου είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, όταν πρόκειται για την προστασία των καταναλωτών, που από τη δική μου τη σκοπιά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, οδηγίας αυτής και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε πού χρειάζονται πρόσθετες πρόνοιες ώστε να λάβουμε υπόψη την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Και υπάρχουν και ορισμένοι συνάδελφοι. Γεια σας. Ίσως λοιπόν αυτός είναι ένας πιο ε, βιώσιμος τρόπος για να λειτουργήσουμε καλύτερα και να υποστηρίξουμε και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για το θέμα της ε, συλλογής δεδομένων, ε, υποστηρίζω αυτό το οποίο είπε η εκθεσή σας για την εισαγωγή μιας κεντρικής τράπεζας δεδομένων και εγώ κατέθεσα μια τροπολογία στο χώρο αυτό, όχι με διαφορετική οδηγογραμμή, αλλά τονίζοντας τη σημασία του να εξετάσουμε πώς θα γίνει αυτή η συλλογή δεδομένων, γιατί είναι σημαντικό και η Κομισιόν να μπορέσει να εξετάσει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων με μια πιο ευρεία αντιμετώπιση και ακολουθώντας μια συνεκτική αντιμετώπιση για το ότι είδου στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα, ποια ελείπουν, ποιος πρέπει να τα, συ... να τα συγκεντρώνει κτλ. ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Αλλά όταν δούμε το εύρυ φάσμα τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια συνισταμένη για όλα αυτά τα θέματα. Στην εισαγωγή σου δεν είδα να υπάρχουν και σχόλια για τις τροπολογίες που θέλουν να υπάρξει μια, ένας διαχωρισμός μεταξύ επενδυτικών τραπεζών και εμπορικών τραπεζών. Τραπεζών δηλαδή με φυσιολογική δραστηριότητα. Θα δείτε λοιπόν ότι η έκθεση της Επιτροπής Λίγκανεν είχε κάνει μερικέ προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια δεν είναι μαύρα ή άσπρα όλα αυτά τα σημεία, αλλά θα ήταν χρήσιμο και η δική μας Επιτροπή να πάρει μια θέση για τον ενδεχόμενο αυτό διαχωρισμό. Και όσο αφορά την αντιμετώπιση των τίτλοποιήσεων, νομίζω ότι πράγματι υπάρχει μια κοινή γραμμή που διατρέχει τις τροπολογίες και η οποία είναι θετική και επίσης για τη ρύθμιση των λεγόμενων ε, money market funds, δηλαδή των ταμείων πρόθεσμων επενδύσεων, θα ήταν χρήσιμο να περιλάβουμε και αυτά στο τα ταμεία στο πλαίσιο ρύθμισης και να ευθυγραμμιστεί η αντιμετώπιση τους με τον τρόπο αυτό. Όταν πρόκειται τώρα για τους ε, δίκτες που ακολουθούν, για, τους, ε, για τα ταμεία που ακολουθούν τους χρηματιστηριακούς δείκτες, τα Exchange Traded Funds, νομίζω ότι και για αυτά τα ταμεία θα πρέπει να υπάρξει μια συμπερίληψη μέσα σε αυτό το πλαίσιο και βλέπω να υπάρχει ήδη κάποια σύγκληση μέσα από τις τροπολογίες και επομένως θα μπορούσαμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Και με όλα αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην ουσία του θέματος. Βλέπουμε που είναι τα προβλήματα και μπορούμε έτσι να δούμε για ποια, πράγματα, για ποια θέματα χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία και φυσικά βασίζει, μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα στην δική μας ε, υποστήριξη και θα αναφερθώ στις τροπολογίες λεπτομερέστερα όταν χρειαστεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αδιαμφισβήτητο είναι για μένα, πιστεύω, ότι ένας από τους λόγους για την παγκόσμια ε, χρηματοπιστωτική κρίση ήταν το λεγόμενο ρυθμιστικό αρμπιτράζ, η επιλογή δηλαδή ρυθμιστικού πλαισίου. και το γεγονός ότι η προσπάθεια να υπάρχει καλύτερη ρύθμιση του πιστοτικού συστήματος, του τραπεζικού και πιστοτικού συστήματος, οδήγησε σε μια έκρηξη του, ε, του ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Επομένως θα πρέπει να ασχοληθούμε και για το θέμα αυτό. Η έννοια σκιώδες τραπεζικό σύστημα είναι λίγο άστοχη, το ξέρουμε όλοι, γιατί κάπου φαίνεται να είναι σκοτεινές ενέργειες, ε, ενέργειες αμφίβολης νομιμότητας κτλ. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, δραστηριότητες οι οποίες είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπορυθμιστικό πλαίσιο, αλλά δεν υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια σε σχέση με αυτές. Εγώ έχω καταθέσει οκτώ τροπολογίες, αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτω τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του Σαϊντ Ελχάντραουι, τις αντιμετωπίζω ιδιαίτερα θετικά και τις υποστηρίζω και νομίζω ότι έχουμε σχεδόν μια συνένεση για τα θέματα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε, θα δυσκολευτούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να δεχτούν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα του τομέα του σκιώδους πιστοτικού συστήματος είναι η έλλειψη διαφάνειας και επαρκής παροχή επαρκούς παροχής πληροφοριών. Γι' αυτό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί με τους εταίρους μας, όπως είναι οι ΗΠΑ, να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει να υπάρχει καλύτερη υποπτία του τομέα αυτού του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Τώρα, το, για το ερώτημα μέχρι πότε θα πρέπει να επιτευχθεί μια ρύθμιση, εγώ θα έβλεπα να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, ίσως υπερβολικά φιλόδοξο, να θεωρήσουμε ότι μέχρι τις αρχές του 2013 θα πρέπει να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ούτε τρεις μήνες δεν μας μένουν για να τα επιτελέσουμε όλα αυτά. Αν μπορέσουμε όμως να επιτύχουμε μέσα στο 2013 να έχουμε μια ρύθμιση, αυτό για μένα μου φαίνεται θετικό. Υπάρχουν ήδη ε, πολλά νομοθετήματα και οδηγίες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα για, τους, ε, για τα ταμεία που βασίζονται σε χρηματοριστιακούς δείκτες, τα exchange traded funds και άλλα τέτοια ε, πιστοτικά μέσα μπορούν να εφαρμοστούν ήδη αυτές οι ρυθμίσεις. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα καλύτερο και νέο ορισμό των επιλέξιμων ε, στοιχείων ενεργητικού, ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα θέματα αυτά και να μπορούμε να ξέρουμε ότι οι εγγύησεις αυτές Επίσης, στις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει πολλές κινήσεις και υπήρξε και επαφή με τους άλλους ε, σκιώδεις Υπήρξε πάρα πολύ θετικό κλίμα για ε, συζήτηση σε σχέση με τα money market funds και υπήρξαν και πολλές συζητήσεις σε πάνελ για τα θέματα αυτά και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ήδη ο ίδιος ο χρηματοπιστωτικός τομέα, οι τράπεζες ιδιαίτερα που ενδιαφέρονται το ταχύτερο δυνατό να γνωρίζουν ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί και ποιε θα είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι δύσκολο όμω ακόμα να καταλήξουμε σε μια σαφή κατεύθυνση για το τι θα κάνουμε ή όχι στην Αμερική. Η εντύπωση ήταν ότι οι ΗΠΑ είχε καταφέρει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να πει στον κύριο Σαπύρο και άλλους ότι δεν, η πρότασή τους δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο κύριος Γκάιτνερ πάντως υποστηρίζει ότι οι προτάσεις αυτές είναι χρήσιμες και πρέπει να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Ευρώπης. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένες και κεφαλοχικής επάρκειας. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν και στα πλαίσια συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις αναφορές και τις εκθέσεις, νομίζω ότι μία ε, έκθεση για την χρηματοπιστωτική κατάσταση και την κατάσταση εποπτείας να δίδεται, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που να κάνουν σαφή την κατάσταση. Επίσης για την αναδιάρθρωση των τραπεζών και επίσης για τα θέματα της τιτλοποίησης ορισμένου στοιχείου ενεργητικού. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες και προδιαγραφές γιατί δεν μπορούμε να πούμε έχουμε τις προτάσεις ήδη για την τιτλοποίηση μπορούμε να πούμε ότι μια τιτλοποίηση μπορεί να εγγράφεται στα λογιστικά στοιχεία μέχρι κάποιο επίπεδο, όχι να αλλάζει συνέχεια το επίπεδο ε, το οποίο εγγράφεται για μια τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού. και για, ε, ε, για τα ομόλογα και για τα ρέπο, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε με τους εμπλεκόμενους στην αγορά αυτή και να τους αφήσουμε αυτοί να αποφασίσουν κάτω από ποιε συνθήκες είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν ένα κούρεμα με σε εισαγωγικά και μέχρι ποιου ύψου μπορεί να φτάσει αυτό το κούρεμα. Εμείς δεν μπορούμε αυτό ως νομοθέτες να το επιβάλλουμε, ούτε να του επιβάλλουμε ποιο θα ήταν το αποδεκτό και το σωστό επίπεδο για ένα κούρεμα. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο είχα ξεχάσει να αναφέρω για τα, για τα μηδέα κεφάλαια χρηματαγοράς, τα money market funds, έχει δείξει η κρίση ότι ακόμα και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς τα οποία βασίζονται σε ισοτιμία δολαρίου δεν έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά οι, αυτοί που χρησιμοποιούν τα αμοιβαία κεφάλαια κεφαλαίου δεν του ενδιαφέρει κυρίω το κέρδο, του ενδιαφέρει η ευκαμψία και η ρευστότητα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα μήπω τα πρώτα δύο σημεία να αναφερθούν στις προδιαγραφές μας. Η εξασφάλιση της ασφάλειας, βέβαια με κάποιο τίμημα, και επίσης η ρευστότητα. Και τώρα, αν είναι οι αμερικάνικες ε, λύσεις, αν θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό των, των ταμείων αυτών που να μπορούν να αναλυφθούν σε ημερήσιο ή σε εβδομαδιαίο επίπεδο, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να, να παραγνωρίσει το γεγονός ότι ενώ φαίνονται απόλυτα ασφαλή τα μηδέα κεφάλαια ε, κεφάλαια χρήματα δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο ασφαλή ούτε τόσο διάφανα. Ξέρουμε ότι σε παραπάνω από μία περίπτωση έχουν βρεθεί σε δυσκολίες και η τράπεζα η οποία είχε ουσιαστικά ε, δημιουργήσει αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια χρειάστηκε να παρέμβει και να διασώσει αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. Είναι πολλές φορές που έχει γίνει αυτό και πριν από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ότι χρειάστηκε να διασωθούν τέτοια αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και αυτό επομένως στο μέλλον θα πρέπει να καλύπτεται με μεγαλύτερη διαφάνεια. Ένα ακόμα ε, κύριο πρόβλημα, ένα κέριο πρόβλημα είναι το θέμα πώς με το χαμηλό επιτόκιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή όταν δεν υπάρχουν ουσιαστικά επιτόκια, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα αμοιβαίο ταμείο χρηματαγοράς, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς όταν δεν υπάρχουν πια οι δυνατότητες κερδοφορίας. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταγράψουμε εμείς στους κανονισμούς και στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Οι τροπολογίε νομίζω ότι είναι πολύ σαφεί, πολύ εύληπτε, αυτονόητε θα έλεγα, ο site. Ναι, μόνο να ευχαριστήσω τους συναδέρφους που πήραν το λόγο. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα. Όπως είπα και στην αρχή, μέσα στις επόμενες ημέρες θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες και έτσι να έχουμε μια καλή πρόταση ώστε να γίνει και η ψηφοφορία απρόσκοπτα μέσα σε μερικές μέρες. Ωραία, ευχαριστώ. Θέλουμε να ψηφίσουμε στις 22 ε, Οκτωβρίου. Είναι εβδομάδα Στρασβούργου αυτή. Έτσι προβλέπεται στο χνοδιάγραμμα. Και σκοπό έχουμε να πάει το θέμα στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ωραία, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είμαστε αρκετά εντάξει με το χρόνο, λίγα λεπτά πιο πριν τελειώσαμε από τι περιμέναμε. Ε, ο Λίαμ είναι εδώ, έρχεται. Ο Βόλφ είναι εδώ, ο Θείοντορ, ο Φίλιπ δεν είναι εδώ, η Εύα είναι εδώ και ο Νίκολας. Σχεδόν είμαστε όλοι εδώ. Μπορούμε να πάμε στο τέταρτο σημείο της ημερησίας διάταξης, που είναι το πρόγραμμα φυσκάλης. Ο Φιοντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι ήδη κάνουμε μια συζήτηση για το πρόγραμμα αυτό. Για πρώτη φορά η Κομισιόν πρότεινε ένα πρόγραμμα που θα ονομαζόταν Φίσκρους ήταν ένα πάντρεμα του περασμένου, του παλιού προγράμματος φισκάλης και του προγράμματος για τα τελωνία. Με βάση την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Κομισιόν αποφάσισε τελικά να επανέλθει με ένα χωριστό πρόγραμμα ή προγράμματα, ένα φισκάλης και ένα χωριστό για τα τελωνία. Είμαστε δηλαδή στο ίδιο πλαίσιο με παλιά, δηλαδή με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Κομισιόν που επανήλθε και υπέβαλε πρόταση με βάση αυτά που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το νέο πρόγραμμα φυσκάλης λοιπόν τώρα, το οποίο έχουμε μπροστά μας και εξετάζουμε, έχει δύο βασικά συστατικά, δύο βασικές συνιστώσεις. Καταρχάς είναι να υποστηρίξει την φορολογική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Και η δεύτερη βασική συνιστόσα του προγράμματος αυτού είναι να υποστηρίξει την ε, προσπάθεια δημιουργίας δυναμικού πληροφορικής, μηχανοργάνωσης. Μιλάμε εδώ για πολλές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των ε, φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Φισκάλης 2007-2013, αξιολογήθηκε από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές. Ο ένας αξιολογητής ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα, την προσθέμενη αξία που προσέφερε το πρόγραμμα αυτό. Και ένας άλλος αξιολογητής ασχολήθηκε με τις δυνατότητες βελτίωσης του μελλοντικού προγράμματος φυσκάλης, δηλαδή 2014-2020. Να τονίσω ότι οι αξιολογητές εκφράστηκαν πολύ θετικά για αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που ανταποκρινόταν, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών έχει σαφή προστιθέμενη αξία γιατί η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών είναι πάρα πολύ σημαντική ούτως ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Επίσης, η Κομισιόν, την οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε, έλαβε υπόψη της όχι μόνο τις συστάσεις του δεύτερου αξιολογητή, ο οποίος αξιολόγησε το πώς μπορεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα φυσκάλης την επόμενη περίοδο, δηλαδή 2014-2020, αλλά έλαβε επίσης υπόψη η Κομισιόν στο νέο πρόγραμμα που μας παρουσίασε. Έλαβε λοιπόν υπόψη και κάποιες από τις δικές μας συστάσεις συστάσεις που είχαν ε, προκύψει από τις συζητήσεις μας. Εστιάζοντας πολύ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και της επιθετικής φόρο αποφυγής. Ε, και αυτό θα πρέπει να το επιτύχουμε χάρη στην στενότερη συνεργασία των φορολογικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το πεδίο εφαρμογή του προγράμματος. Η πιο σημαντική βελτίωση είναι η πρόταση της Κομισιόν να μην περιοριστεί το πρόγραμμα μόνο στο ΦΠΑ, στις, στους ειδικού φόρους κατανάλωσης, στην άμεση φορολογία, αλλά και σε άλλους φόρους που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Φορολογική Νομοθεσία. Φερρυπίν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε υιοθετήσει κανονισμούς για την ανάκτηση χρεών μέσω της συνεργασίας των φορολογικών αρχών των χωρών μελών. Επίσης υπάρχει μια πρόταση σε αυτή τη συνεργασία για συμμετοχή και των υποψηφίων χωρών, δυνητικών υποψηφίων χωρών και χωρών της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας υπό κάποιες προποθέσεις όμως. Επίσης η Κομισιόν πρότεινε να συμμετάσχουν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες, από τα Υπουργεία Οικονομικών κτλ αλλά και από διεθνείς οργανώσεις. Όπως είπα, οι συστάσεις μας από την προηγούμενη συζήτηση ήταν να υπάρχουν σαφείς προτεραιότητες ε, κατά της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης, καθώς και η μείωση του διοικητικού άχθους που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Το πόσο που διαθέτει το πρόγραμμα αυτό είναι 234 εκατομμύρια ευρώ για όλη την περίοδο 2014-2020. Έχουμε μια τροπολογία εδώ, που είναι κοινή για τέτοιου τύπου προγράμματα, ότι αυτό το ποσό δεν είναι το τελικό, γιατί πρέπει να περάσει πρώτα από τις τελικές διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε για το πολιτευσιμο οικονομικο οικονομικό πλαίσιο 2014-2020 και εκεί θα αποφασιστεί ποιο θα είναι το τελικό ποσό. Αυτό προτείνουμε στις τροπολογίες μας, στο σχέδιο κανονισμού. Καταρχάς, προτείναμε να εστιάσουμε στη συνεργασία με ενδεχόμενες υποψήφιες χώρες και με χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και η συνεργασία αυτή να έχει σαν στόχο την καταπολέμηση φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει περιορισμένους πόρους. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων υπαλλήλων τρίτων χωρών, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων, προτείνουμε μια περιορισμένη εμπλοκή και συμμετοχή τέτοιων ε, εμπειρογνωμόνων, γιατί ακριβώς έχουμε περιορισμούς οικονομικούς. Έχουμε λίγους πόρους στη διάθεσή μας στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, Υπάρχει μια τροπολογία και θέλουμε να πετύχω μέσω αυτής το να μην χρησιμοποιηθούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διμερή συνεργασία μεταξύ μιας ενωσιακής χώρας και μιας τρίτης χώρας, να μην χαθούν αυτά τα λεφτά, γιατί η Κομισιόν πρότεινε μέσω αυτού του προγράμματος να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε να έχουμε συνεργασία μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας ή δύο τριών, τρίτων χωρών, ε, θέματα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω διμερών σχέσεων. Γι' αυτό λοιπόν προ, προτείναμε τέτοιες τροπολογίες, ούτω ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη και τουλάχιστον τρίτες, ε, και τουλαχιστον τουλάχιστον δύο και τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες σε αυτή τη συνεργασία. Μια άλλη τροπολογία, Και τη συζητήσαμε πολύ με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Υπάρχει μια ανακοίνωση που λάβαμε από τον πρόεδρο Μπαρόζο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο πρόεδρος συστήνει να μην έχουμε ανώτατα όρια μέσα στο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν ανώτατα όρια, έτσι όπως το προτείνει η Κομισιόν. Γιατί τα ανώτατα όρια περιορίζουν την ε, δυνατότητα εφαρμογής που έχει η Κομισιόν στη φάση εφαρμογής. Η σκέψη μας ήταν η εξή. Το πρόγραμμα έχει δύο βασικές ε, συνιστώσεις. Συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών, δηλαδή κατάρτιση, σεμινάρια, διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπου οι φορολογικές αρχές ανταλλάσσουν και γνώσεις και καλές πρακτικές και δυνατότητα οικοδόμησης ε, δυναμικού ε, πληροφορικής. Και με βάση την εμπειρία που έχουμε από το προηγούμενο πρόγραμμα 2007-2013, τα περισσότερα χρήματα από αυτό το πρόγραμμα πηγαίνουν τελικά στην ε, προσπάθεια οικοδόμησης δυναμικού πληροφορικής. Και έτσι ανταλλάσσουμε πληροφορίες αυτόματα για το ΦΠΑ, για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Εμείς είπαμε ότι μπορούμε να ξοδέψουμε μέχρι τόσα για την οικοδόμηση πληροφορικής και είπαμε ότι το πολύ πολύ το 80% των πόρων θα πάνε για την πληροφορική ούτως ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του τομέα αυτού της πληροφορικής και της συνεργασίας των φορολογικών αρχών. Επίσης, υποβάλα μία τροπολογία, ούτως ώστε οι εκθέσεις για τις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις και η τελική αξιολόγηση να αποστέλλονται επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε σαφέστερη εικόνα και να υπάρχει λογοδοσία από πλευράς της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Αυτά είχα να πω. Α δούμε τι έχουν να πούν οι σκιώδει ηγητέ, α δούμε τι έχουν να πούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και βεβαίω και ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ο κ. Δασκάλου, που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή. Αν έχουμε χρόνο, η Επιτροπή στο τέλο θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Στόλογιαν. Λέει η κυρία Φερέρα. Η Λίνα δεν μπορούσε να είναι εδώ. Είχε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση στη χώρα του και μου ζήτησε εγώ να τον αντικαταστήσω και να μιλήσω εκ μέρους του. Είχε την ευκαιρία, έτσι αλλιώ, ήδη από τον Ιούνιο να ευχαριστήσει τον κύριο Στόλογιαν για την πρώτη του έκθεση όσον αφορά το φισκάλις. Τώρα θέλει να ευχαριστήσει και πάλι για τη δεύτερη αυτή έκθεση. Και εκείνος και εγώ με ικανοποίηση βλέπουμε ότι η Επιτροπή επιτέλους προτείνει τροποποιημένη πρόταση από τον Αύγουστο. Ε, το μόνο το οποίο δεν μας ικανοποιεί είναι το ότι δεν έγινε αυτό νωρίτερα. Υπάρχουν έτσι καθυστερήσεις, μεγάλος φόρτος εργασίας για όλους. Έρχομαι τώρα στο νέο σχέδιο έκθεσης. Πολλοί είναι πιστεύει, καλά έτσι καλώς δεν χρειάζεται να επαναλάβω τώρα ότι έχουμε ήδη πει τον Ιούνιο, αλλά υπενθυμίζει ότι Κύριε Σιγητά, συμφωνούμε μαζί σας όσον αφορά την ενίσχυση ε, του προγράμματος, ώστε αυτό να επικεντρώνεται στην φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Το είναι πάρα πολύ και την φοροαποφυγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για όλους εδώ στην Επιτροπή μας. Όμως, δεν αναφέρεστε στη διπλή φορολόγηση ή στη διπλή μη φορολόγηση, στην προηγούμενη τροπολογία αριθμός 8 που τώρα είναι η τροπολογία 5. Η διατύπωση αυτή ευθυγραμμιζόταν και με τη δουλειά που είχε κάνει η Επιτροπή μας στον τομέα της φορολόγησης πρόσφατα. Τώρα για τις άλλες τροπολογίες υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο δεύτερο αυτό σχέδιο, αν το συγκρίνουμε με το πρώτο. Για παράδειγμα, με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τροπολογία 9, η διατύπωση εδώ επιτρέπει, πιστεύω, έναν, και ο κύριος Λίνε, δηλαδή πιστεύει, μια καλή συμβιβαστική λύση. Σημειώνει επίσης ο συνάδελφος ότι φύγαν οι οροφές που είχατε στην πρώτη έκθεση για τις διάφορες επιλεγμένες δράσεις, το τέος άρθρο 6 και το ρινό άρθρο 7. Τα επίπεδα όμως οροφής θα πρέπει να συζητηθούν με τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πεπισμένος ότι οι οροφές στον κανονισμό θα βοηθούσαν να ελέγξουμε καλύτερα την ε, εκτέλεση του προγράμματος. Τέλος, όσον αφορά για τις κοινέ δράσεις και τους πολύπλευρους ελέγχους έχετε εισαγάγει στο δεύτερο σχέδιο πιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να επιλέγονται τέτοιες δράσεις. Λέτε ότι θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον τρεις χώρες, δύο από τις οποίες να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λίμι θα ήθελε να καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή τώρα. Κατά τη γνώμη του, η ευρωπαϊκή διάσταση διασφαλίζεται και με ένα ελάχιστο δύο χωρών μελών. Εμείς θα ετοιμάσουμε τροπολογίες που ελπίζουμε να βρείτε επικοδομητικές και όλοι είναι περιμένει καρποφόρα συνεργασία μαζί σας. Προβλέπει σε αυτήν και σας ευχαριστώ όπως επίσης και εγώ για την δουλειά σας μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Ο Βόλφ. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά γιατί μετά από αυτά τα οποία είπε και ο εισηγητής και οι υπόλοιποι εισηγητές δεν μένουν πολλά πράγματα στον κατάλογό μου. Μπορούμε να πούμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πράγματι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια θετική ενέργεια λοιπόν από την πλευρά της Κομισιόν και αποτελεί μια καλή βάση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο εισηγητής έχει καταθέσει μονάχα ένα περιορισμένο αριθμό τροπολογιών και τώρα και αυτό αντικατοπτρίζει και την ποιότητα της προτάσης της Κομισιόν. Έρχομαι τώρα σε πιο λεπτομεριακά θέματα. Ένα ερώτημα είναι ποιος θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε τέτοια προγράμματα. Φαίνεται ότι και η Κομισιόν και ο εισηγητής πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει περιορισμένη η συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Αλλά ο ορισμός αυτός ο οποίος έχει προταθεί από τον εισηγητή μπορεί να γίνει σαφέστερος σε σχέση με τους εμπειρογνώμονες. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εδώ θέλουμε να έχουμε εμπειρογνωμοσύνη μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο για να φέρουμε σε πέρα στον συγκεκριμένο στόχο που έχουμε. Αν δηλαδή φαίνεται ότι με τη συμμετοχή αυτών των εμπειρογνωμών θα μπορέσει να υπάρξει μια ορατή βελτίωση στην ε, αντιμετώπιση της φοροαπάτης και της φοροαποφυγής. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, εγώ κατανοώ ότι λέει ο εισηγητής ότι δεν θα πρέπει να δαπανίσουμε το σύνολο αυτών των κονδυλίων για την ε, <clears throat> ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Αν το 80% που προβλέπει αυτός για την πρόληψη είναι το καλύτερο ποσοστό ή όχι, εμείς πάντως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα προγράμματα να είναι τόσο καλά επιλεγμένοι και τόσο καλά ε, εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά αυτά τα δύο προγράμματα. Αυτό μου φαίνεται εμένα ότι είναι το πιο σημαντικό. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μια διαφορετική κατανομή κονδυλίων από το 80-20% που προτείνει ο εισηγητής και εξάλλου υπάρχει μια τεράστια πολυπικιλία σε σχέση με το επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων στα τομέα, στον τομέα αυτό μεταξύ των διαφορών κρατών μελών. Μπορεί χωρίς τώρα να σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά υπάρχει ένα κράτος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, αποτελεσματικότητα της δίκησης. Μπορεί πραγματικά να είναι διαφορετική λοιπόν η κατάσταση σε μια χώρα από τη στην σε ό,τι αφορά το επίπεδο κατάρτισης των ε, υπαλλήλων στα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο επομένως να εξασφαλίσουμε ότι με ανάλογες ενέργειες καταρτήσεως θα φτάσουμε σε ένα κοινό επίπεδο ε, κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το 80% που προτείνει ο συγητής. Τρίτο σημείο. Βέβαια πρέπει να καταμετρήσουμε και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών αν δεν είναι αποτελεσματικά δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τέτοια προγράμματα. Αλλά απλώς μου φαίνεται ότι οι προθεσμίες που προτείνει ο εισηγητής για την ενδιάμεση ε, αντιμετώπιση και την τελική ε, έκθεση δεν είναι επαρκή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο να γίνεται μια τακτική επισκόπηση για να είμαστε σίγουροι <clears throat> ότι επιτυγχάνουμε την πρόοδο όπως προτείνεται από την Κομισιόν και σας υπενθυμίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια λέμε ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεπεράσουν τις αναποτελεσματικότητες στη συλλογή των ε, φορολογικών εσόδων. Και επίσης να αντιμετωπιστεί καλύτερα η, η φοροαποφυγή και η φοροαπάτη και δεν έχουμε πετύχει τίποτα στον τομέα αυτό. Βλέπουμε να υπάρχει το ίδιο αν όχι και μεγαλύτερο επίπεδο φοροαπάτη στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και αυτό είναι ακόμα πιο οξύ σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και γι' αυτό για μένα το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε 32 εκατομμύρια ή περισσότερα ή λιγότερα εκατομμύρια. Το θέμα είναι να δώσουμε τους απαραίτητους πόρους ώστε σε τελική ανάλυση να μπορέσουμε να έχουμε την πρόοδο η οποία θα είναι απτή και ορατή και για τον πολίτη στην καταπολέμηση της φοροαπάτησης και φοροαποφύγης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ εύγλωτη εξήγηση και παρουσίαση της πρότασης. Έχω σκεφτεί μερικές παρατηρήσεις. Καθώς τις ξαναβλέπω, βλέπω ότι ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτά που είπαν ο κύριος Στολογιάν και ο κύριος Κλίντ. Ούτως ώστε οι δαπάνες που θα κάνουμε να αποδώσουν. Ένα γενικό σχόλιο θα ήθελα να κάνω καταρχήν. Ο κύριος Τολογιάν ανέφερε στην ομιλία του την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που μπορεί να οδηγήσει σε επίταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας είναι το κράτος δικαίου να λειτουργεί και στις φορολογικές αρχές και η δική μου πολιτική ομάδα συμφωνεί απόλυτα με την έκθεση αυτή, η ομάδα των συντηρητικών. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Στολογιάν που ζητάει αποτελεσματική και έντονη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών. Όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής. Και τονίζει ποιες είναι αυτές οι τρίτες χώρες που μπορούν να συνεισφέρουν, να συμμετέχουν είναι είτε υποψήφιες χώρες, είτε πιθανές υποψήφιες χώρες. Επίσης, συμφωνώ με την ε, στενότερη συνεργασία των φορολογικών αρχών με σκοπό να περιοριστούν ουσιαστικά οι φορολογικές απάτες και η φοροδιαφυγή. Πώς να διαφωνήσουμε με αυτό. Τώρα είμαστε πιο προσεκτικοί, όμως, σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε απόπειρα, να ενισχύσουμε την φορολογική εναρμόνιση, που είναι η τροπολογία υπαριθμών 3, ή να θέσουμε ελάχιστα φορολογικά όρια. Θα συζητήσουμε αυτή την τροπολογία με τον εισηγητή θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Το Φισκάλις και άλλα προγράμματα αντίστοιχα στο μέλλον, κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν παιχνίδια εναρμόνισης που σκοπό θα έχουν να εναρμονίσουν την το επίπεδο φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτές οι αποφάσεις είναι δουλειά των κρατών μελών. Και θα πρέπει, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν σε επαφή και σε διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για να επιλύνουν τα διμερεί προβλήματα. Επίσης, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, ναι, συγκεκριμένοι όμως και επιλεγμένοι. Να υπάρχει ένα κατάλογος επιλεγμένων ε, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων αν θέλουμε να προσλάβουμε αρχαίο εμπειρογνώμονα, θα πρέπει να είναι ο καλύτερο. Και αντίστοιχη πληρωμή, βέβαια, να προβλέψουμε αυτού του ανθρώπου. Όλη η διαδικασία επιλογής αυτών των ε, εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να είναι διαφανής. Προφανώς δημόσια σημαίνει αυτό. Επίση, για τα λεφτά. Τι να πω παραπάνω από αυτά που είπε ο κύριος Κλίντ. Συμφωνώ απόλυτα. Προσοχή. Δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύουμε χρήματα για φανταχτέρη πληροφορική. Θα πρέπει να επενδύουμε χρήματα για κατάρτιση, για υποστήριξη και προώθηση της συνεργασίας, των βέλτιστων πρακτικών. Αυτές είναι οι τροπολογίες μου. Ετοίμασα μια ομάδα τροπολογιών και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία πολεμική γύρω από αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, Νίκολας. Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την παρουσίαση που έκανε και ειδικά έτσι όπως μας εξιστόρισε το ιστορικό αυτής της υπόθεσης ε, να τον ευχαριστήσω από το γεγονός ότι με τις προσπάθειες της δικές του και της Επιτροπής, επιτέλους, της Επιτροπής μας και άλλο, επιτέλους η Κομισιόν κατάλαβε ότι πρέπει να ξεχωρίσει τα δύο αυτά προγράμματα, δηλαδή της φορολογικής α, συνεργασίας και το θέμα των τελωνίων και έτσι μπορούμε να δουλέψουμε αποτελεσματικά στο ένα το συγκεκριμένο που συζητάμε τώρα και που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης. Η δεύτερη μου, οι παρατηρήσεις μου από εδώ και πέρα έχουν το χαρακτήρα ότι ενδεχομένως κάποιες τροπολογίες που θα καταθέσουμε θα είναι στο πνεύμα που θα αναφέρω εδώ και θα είμαι σύντομο. Οπωσδήποτε χρειάζεται συνεργασία των φορολογικών δικήσεων των κρατών μελών για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη τα πληροφοριακά συστήματα είναι βοηθητικά και απαραίτητα, αλλά θέλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αυτή η πλευρά είναι η τεχνική πλευρά της υπόθεσης. Η πολιτική και η ουσιαστική πλευρά είναι ποιον κυνηγάμε, ποια φοροδιαφυγή θέλουμε να συλλάβουμε. Και εδώ είναι φανερό και είναι μια πολιτική παρατήρηση ότι δεν υπάρχει ισχυρότατη βούληση και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη στο να αντιμετωπίσουν τους επαγγελματίες μεγαλοφοροφυγάδες. Αναφέρομαι της χάρη στις πολυεθνικές που φοροδιαφεύγουν ανενόχλητες καθώς μεταχειρίζονται τις ενδοομιλικές συναλλαγές μεταφέροντας από τις θηγατρικές σε χώρες που έχουν καλύτερο φορολογικό καθεστώς. Και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή. Επομένως, γενικώ η παρατήρηση είναι ότι αυτά τα συστήματα ναι είναι αποτελεσματικά κατά τη γνώμη μου εφόσον έχουν και συγκεκριμένη τέτοια πολιτική στόχευση τόσο ώστε να πάμε σε ένα φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο αναδιαμενεμητικό και αναπτυξιακό. Τέλος, η τελευταία μου παρατήρηση είμαι πιο, ε, θα σας έλεγα, πιο επιφυλακτικός ακόμα και με αυτή την προσεκτική τοποθέτηση που κάνει ο εισηγητής μας σχετικά με τον περιορισμένο, περιορισμένη ε, αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων, η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζονται εμπειρογνώμονες για να μπορέσει να υπάρξει μια ε, συνεργασία καλύτερη μεταξύ των εθνικών φορολογικών δικήσεων, πολύ δε περισσότερο που παρά την, ας το πούμε έτσι, κάποια περιγραφή, υπάρχει μια σάφια περί τίνος πρόκειται ποιοι θα είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονε και γιατί δεν του διαθέτει ας πούμε, τα κράτη για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Επομένω, καταρχήν λέω δεν συμφωνώ, δεν συμφωνούμε με την αναγκαιότητα συμμετοχή στο πρόγραμμα ξένων εμπειρογνωμόνων. Αυτέ είναι οι βασικέ μα παρατηρήσει και στο πνεύμα αυτό ενδεχομένω θα καταθέσουμε κάποιε τροπολογίε. Κατά τα άλλα ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Um, Έχουμε χρόνο να λάβει το λόγο η Κομισιόν εφόσον το επιθυμεί. Thank you very much, Madam Chair. Μερσή, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ταχεία διεκπαιρέωση της πρότασής μας και την πολύ καλή του έκθεση. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο γιατί με τρόπο εντελεχή έχει εξηγήσει αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση Φισκάλης 2020. Κάποια σχόλια έχω να κάνω μονάχα σε σχέση με την, με την δική του πρόταση και αυτά που ανέφερε ο κύριος Κλίντς. Για τον εισηγητή και την πρότασή του θέλω να κάνω κάποιες ε, επιφυλάξεις για τροπολογία 30 που αφορά τον πολυμερή έλεγχο. Πιστεύουμε ότι το τωρινό κείμενο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την νομοθεσία για τη διοικητική συνεργασία και ο πολυμερής έλεγχος όταν ασκείται από δύο χώρες παραγωγής χάρη δείχνει ότι δεν δημιουργεί προβλήματα και δεν εμποδίζει την σωστή εφαρμογή. Και αυτό περιλαμβάνεται τώρα στο πρόγραμμα φυσκάλης. Η δεύτερη επιφύλαξή μου αφορά την τροπολογία υπαριθμών 15 και άπτεται της, του ορισμού μιας οροφής που να είναι 80% σε σχέση με... Όχι, δεν είναι στο σημείο. Στην τροπολογία 15, μια στιγμή. Είναι τροπολογία 14, συγγνώμη. Όπου προτείνεται να υπάρξει οροφή σε σχέση με το τμήμα των κονδυλίων που αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση σε πληροφοριακά συστήματα στο 80% μονάχα. Για μας αυτό ε, υποσκάπτει λιγάκι την ευελιξία η οποία προβλέπει το πρόγραμμά μας και πιστεύουμε ότι σε μια ενδιάμεση αξιολόγηση θα έχουμε τη δυνατότητα ήδη μέσα στην ε, ζωή του προγράμματος αυτού που θα κρατήσει 7 χρόνια να αλλάξουμε την κατανομή των πόρων του προπολογισμού επί τη βάση των αναγκών. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα χρειαστούν τα χρήματα αυτά και θα ήταν πραγματικά πιο αποτελεσματικό να έχουμε πλήρη ευελιξία σε, στην κατανομή των κονδυλίων και με τρόπο ο οποίο θα είναι διάφανο γιατί γίνεται αυτό επί τη βάση ετησίων προγραμμάτων. Θα θέλαμε όμω να διατηρήσουμε την ευελιξία στον τομέα αυτό. Για τα σχόλια τώρα του κυρίου Κλίντ, θέλω να σα δώσω δύο πληροφορίε. Πρώτα απ' όλα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του σχεδίου πρότασής μας, η κατάρτιση υπόκειται στην εθνική αρμοδιότητα. Η κατάρτιση αυτή και η δημιουργία ικανοτήτων κατά κύριο λόγο γίνεται από τις εθνικές αρχές. Περισσότερες χώρες έχουν σχολές για τα φορολογικά θέματα που είναι πολύ αποτελεσματικές. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να προσθέσουμε είναι περιορισμένο σε σχέση με το έργο των 27 φορολογικών αρχών στα κράτη-μέλη. Όταν υπάρχει μία ανάγκη και μία, ε, μία ρύθμιση νομοθετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσθέσουμε και ένα πρόσθετο κομμάτι εκπαίδευσης πέραν αυτού που παρέχεται στα κράτη-μέλη. Έχουμε στο πρόγραμμα το τωρινό κάποιες τέτοιες ενέργειες κατά και θέλουμε να τις διατηρήσουμε και να τις συνεχίσουμε γιατί η αντίδραση που είχαμε από τις Εθνικές Φορολογικές Αρχές ήταν πάρα πολύ θετική για τα προγράμματα αυτά. Επίσης θα υπενθυμίσω στον κύριο Κλίντς το άρθρο 16 σε σχέση με την εποπτεία. Στην τρέχουσα πρόταση εμείς προ... προτείνουμε να υπάρξει συνεχής εποπτεία και παρακολούθηση <clears throat> των επιτευμάτων του προγράμματος ώστε να μπορούμε να δίδουμε ε, εκθέσεις σε όλες τις επιλέξιμες δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο αυτό, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα αυτό θα μπορεί να έχει στα χέρια του την, ε, τις πληροφορίες εγκαίρως. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω και σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Uh, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κύριο Στολογιάν και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που έλαβαν το λόγο για τις ε, συστάσεις τους και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί τους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη διατύπωση για ορισμένε από τις τροπολογίες, συμφωνώ απόλυτα. ότι η τροπολογία που την ε, προστιθέμενη αξία από την συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων. Ίσως εδώ μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη συμβιβαστική λύση που θα καλύψει αυτό το σημείο. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είχα και κάποιες συζητήσεις με εκπροσώπους φορολογικών αρχών από διάφορα κράτη-μέλη. Και αυτό μπορεί να είναι μονάχα ένα από τα προγράμματα βάσει των οποίων εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών, όχι στο το επίπεδο αλλά σε μεσαίο επίπεδο μπορούν να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές. Αυτή τη στιγμή μια τέτοια δραστηριότητα ε, που να εξασφαλίσει τη συνεργασία των ε, εκπροσώπων φορολογικών αρχών σε μεσαίο επίπεδο, δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα αυτού του είδους. Εγώ προσωπικά είχα και κάποια εμπειρία σε σχέση με τα πληροφορικά συστήματα στη χώρα μου, σε, με διαφορετικές ιδιότητες και μπορώ να σας πω, πιστεύω, ότι δεν υπάρχει όριο στις αιτήσει για υλικό και χρηματοδότηση σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα. Γι' αυτό εγώ έθεσα αυτό το όριο ότι 80% του προϋπολογισμού, το maximum, θα πρέπει να αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο τεχνολογιών, πληροφόρησης και επικοινωνίας. Και όταν λέμε για το μέγιστο ποσό, λαμβάνουμε υπόψη και την πρακτική που ακολουθήθηκε στη διάρκεια του φισκάλης 2007-2013. Έχω διαβάσει βέβαια και την ε, ανακοίνωση του κυρίου Μπαρόζου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, που αφορά την ανάγκη για μεγαλύτερη ευκαμψία. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πετύχει κάποια πρόοδο. Είχαμε περισσότερες επιμέρους οροφές στις προηγούμενες εκθέσεις. Τώρα έχω μονάχα μία οροφή για να μπορέσουμε να, να διαχωρίσουμε τα κονδύλια που πηγαίνουν για την πληροφορική και αυτά που πηγαίνουν για λειτουργικές ενέργειες και ανταλλαγή απόψεων και των πρακτικών. Βέβαια, αυτό θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε μεταξύ των σχεδόν εισηγητών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των άλλων συναδέλφων και πιστεύω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμφωνία στον ε, τριμερή διάλογο αν παραμείνουμε στα πλαίσια αυτής της ε, πρότασης. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσουμε να περατώσουμε το ταχύτερο δυνατό αυτή την ε, έκθεση και απλώς να σας πω ποια είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι εξέταση τροπολογιών 5 ή 6 Νοεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 28 και 29 ή 29 Νοεμβρίου. και διακόπτω την συνεδρίαση μέχρι τις 4.30 όταν θα αφηχθεί ο Επίτροπος Αλμούνια για μια ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική ανταγωνισμού. Right. Um, Καλώς ήρθατε. Κύριε Αλμούνια, στην Επιτροπή μας. Ως ήθιστε, ο Επίτροπος θα μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Θα πάρει πρώτος το λόγο και μετά ο εισηγητής Σάντσεφ πρεσάδο θα πάρει το λόγο μετά η Σκιώδης και μετά όποιος άλλος θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ, κύριε Αλμούνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε και που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα σας παρουσιάσω τα κύρια στοιχεία του προγράμματος εργασίας μας για του χρόνου όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Ίσως κάποια από εσά να διαπιστώσατε ότι στις πρόσφατες παρουσιάσεις μου προσπάθησα να διευκρινίσω τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες, στα διάφορα μέσα για τα, τον ανταγωνισμό, είτε πρόκειται για συγχωνεύσεις, είτε πρόκειται για ελέγχου από το κράτος κτλ που είναι προτεραιότητες με άλλες προτεραιότητες που είναι η ανάπτυξη και μια καλή βάση για να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη είναι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Οι πρωτοβουλίες που σας προτείνω σήμερα εμπνέονται ακριβώς από αυτές τις σκέψεις. Προσπαθώ να βελτιώσω αυτό που θεωρώ ήδη ένα πάρα πολύ καλό σύστημα πλαισίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Αλλά καθημερινά αναρωτιέμαι πώς μπορώ να ανταποκριθώ καλύτερα στις τρέχουσες προκλήσεις χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται με το πλαίσιο εξυγχρονισμού και μετά θα αναφερθώ λιγάκι στις δράσεις αντιτράστ. Όπως έχω πει ήδη, στην πρόσφατη ακρόαση με την Task Force υπό το Σάντσες Πρεσέδο, την, η ανακοίνωση που εγκρίναμε τον Μάιο που μας πέρασε, ε, μιλάει για τρεις στόχους. Πρώτον, διασφάλιση των κανόνων, κρατικών κανόνων, οι οποίοι πρέπει να ενισχύουν την ανάπτυξη, έτσι όπως ορίζεται στους στόχους μας για την στρατηγική 2020. Δεύτερον, να υπάρχει εξυγχρονισμός ε, με προτεραιότητες και ενίσχυση δράσεων που επηρεάζουν θετικά την εσωτερική αγορά. Και τρίτον, ε, θέλω να αναφερθώ λιγάκι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία μας με τους τρεις αυτούς στόχους είναι ό,τι καλύτερο στους καιρούς τους σημερινούς όπου θέλουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και συγχρόνως γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για πολλές χώρες μέλη μας να τα καταφέρουν να βρουν δημόσιους πόρους επειδή έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε στρατηγικές προγραμμάτων λιτότητας. Οι δυσκολίες ε, αυτές, δημοσιονομικές, προσθέτουν ένα στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω, που είναι η δυνατότητα ε, δαπάνηση σπόρων από τα κράτη-μέλη μας που δεν είναι ίδια μεταξύ όλων. Όχι μόνο είναι δύσκολο να βρεθούν δημόσιοι πόροι για να χρηματοδοτήσουν όλους τους στόχους της πολιτικής μας και όλα τα μέση, αλλά επιπλέον δεν υπάρχει ισότιμη κατανομή μέσα στην εσωτερική αγορά. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό για μας να διασφαλίσουμε τον κατάλληλο έλεγχο. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Όπως είπα και νωρίτερα, μίλησα με το Κοινοβούλιο, τα... άκουσα τα θέματα που μου θέσατε εσείς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια αποτελεσματική κρατική ενίσχυση, μια καλή δηλαδή κρατική ενίσχυση, με έλεγχο βέβαια επιδοτήσεων και καλά κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Μια κακή, μια στραβή κρατική επιχορήγηση, τότε αυτό που κάνει είναι ότι κάνει τις επιχειρήσεις να μην είναι βιώσιμες στην αγορά. Εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με τη μεταρρύθμιση για την κρατική ενίσχυση θα περιορίσει την ε, δράση που πλήττει τον ανταγωνισμό και θέλω να αναφερθώ και σε κάποιες διαδικαστικές τροποποίησεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις και να επικεντρωθούμε σε δράσεις οι οποίες θα έχουν πιο μεγάλο αντίκτυπο. Πού βρισκόμαστε σήμερα, αφού δηλαδή οθετήσαμε τη στρατηγική αυτή. Κοιτάμε τις διάφορες πρωτοβουλίες και να δούμε πώς θα τις μετατρέψουμε σε κατευθυντήριες γραμμές. Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν και για τις κατευθύνες γραμμές για τις τράπεζες, για τις εξαιρέσεις που πρέπει να τροποποιηθούν και σε διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Συνεχίζεται δουλειά βέβαια για την αναθεώρηση των διαφόρων κατευθυντηρίων γραμμών, για παράδειγμα για τα αεροδρόμια και την αυσιπλοεία, για την περιφερειακή ενίσχυση, για την ε, βιομηχανία, για ε, κεφάλαια κινδύνου, στήριξη του περιβάλλοντος, έρευνα και καινοτομία. Η αξιολόγηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ήταν το πρώτο. Στη συνέχεια περνάμε στη μεθοδολογία. Ο στόχος μας είναι η Ευρώπη να έχει ένα καθεστώς το οποίο να εγκρίνει την κρατική στήριξη όταν διαπιστώνεται κάποια αποτυχία στην αγορά και η στήριξη αυτή να αποτελεί ένα στοιχείο όθησης. Να μειωθεί η γραφειοκρατία και γι' αυτό θέλουμε να επεκτείνουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν τις εξαιρέσεις και θέλουμε να επεκτείνουμε και την ε, βοήθεια που έχει να κάνει με αυτές τις εξαιρέσεις ώστε να βοηθήσουμε την καινοτομία, να βοηθήσουμε σε περίπτωση που υπάρχουν φυσικές καταστροφές ή για ορισμένε περιπτώσεις ε, υποδομών ή για περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών και τέλος για βοήθεια στη δοσοκομεία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει βέβαια να δείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, όπως έχουν ήδη, και να δείξουν πώς καλύπτουν ε, βάσει του κανονισμού αυτού των ε, μαζικών ε, εξαιρέσεων, πώς τα βγάζουν πέρα και πώς δαπανούν το δημόσιο χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τις αποκλειστικές της ευθύνες όσον αφορά την ε, τήρηση των ρυθμίσεων. Το βέβαιο είναι πάντως ότι δεν θα συμβεί όπως συμβαίνει μερικές φορές. Θα αφήσουμε τα κράτη-μέλη να σέρνονται και να μην ε, τηρούν ε, τις ρυθμίσεις. Και τέλος για τα διαδικαστικά θέλω να υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει έρευνες ανατομέα όσον αφορά τον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και να μπορεί έτσι να παίρνει πληροφορίες κατευθείαν από την αγορά. Η δουλειά προχωράει καλά. Δεν είναι μια εύκολη συζήτηση αυτή που κάνουμε. Οι πρώτες επαφές που έχουμε με τα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτή την δυνατότητα να μπορούμε δηλαδή απευθείας να ζητούμε από όσους συμμετέχουν στην αγορά να μας πούν τι γίνεται με τις κρατικές ενισχύσεις για να είμαι ειλικρινής μαζί σας ε, δεν ε, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής ελπίζω όμως ότι θα μπορέσω να πείσω τα κράτη-μέλη ότι είναι θετικό για αυτά όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα αλλά και για τα ίδια τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιείται αυτό ο νέος μηχανισμός όταν μπορούμε δηλαδή να ζητάμε πληροφορίες απευθείας από διάφορους παράγοντες της αγορές και ότι αυτό θα βοηθήσει και τα κράτη-μέλη γιατί θα αντιμετωπίζουμε έτσι λιγότερες δυσκολίες να κάνουμε τη δουλειά μας. Έρχομαι τώρα στην άλλη μου που έχει να κάνει με το αντιτράστη, με τις συγχωνεύσεις και τα καρτέλ. Εδώ πολύ σύντομα να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Στον τομέα της ενέργειας. Πρόσφατα ανοίξαμε τις ε, διαδικασίες κατά της Gazprom για καταχρήσεις όσον αφορά τη, τους ελέγχους. Στη, στον τομέα της πληροφορικής επίσης, με το Google συνεχίζουμε να δουλεύουμε και ε, αναφερούμε και την υπόθεση της Microsoft για να επανέλθουμε στις δεσμεύσεις του 2009 και θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάρουμε κάποια απόφαση από αυτού. Επίσης ε, κοιτάμε και τα θέματα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο είδου πόλεμος ευρεσιτεχνιών και εδώ έχουμε ξεκινήσει έρευνες για την περίπτωση Apple Samsung και για την περίπτωση Microsoft ε, ή Apple κατά της Motorola. Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της πληροφορικής λοιπόν και σε νέους τομείς. Στον τομέα των ηλεκτρονικών βιβλίων για παράδειγμα, όπου και εδώ εξετάζουμε τις ε, υποχρώσεις που αναλαμβάνουν ε, μεγάλες εταιρείες, η Apple για παράδειγμα και στον τομέα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην Universal και την MI υπήρξε μια συμφωνία την οποία εμείς ε, εγκρίναμε στον τομέα της μουσικής με ένα πακέτο το οποίο μας επιτρέπει να ελέγχουμε τέτοιου είδους συγχωνεύσεις. Η ανησυχία μας όταν αναλύσαμε την συγχώνευση αυτή είχε να κάνει με τη νέα ψηφιακή αγορά για τη μουσική. Οι προκλήσεις είναι πολλές γιατί όλα αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ο κλάδος ε, αλλάζει πολύ και πολύ γρήγορα και αυτό εμεί που θέλουμε είναι οι αγορέ να μένουν ανοιχτέ και να υπάρχει ανταγωνισμό. Στο τομέα των τηλεπικοινωνιών τώρα, και εδώ υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις στην ελευθέρωση των αγορών σε μερικές φορές τις περιπτώσεις της Τελεφώνικα και της Τέλεκομ για παράδειγμα ή της ε, Σλοβακικής και της Γερμανικής ε, αντίστοιχης εταιρεία. Κοιτάμε και την πρόταση ανάμεσα στη Χάτσον της Αυστρίας και την Orange της Αυστρίας για συγχώνευση. Και έχουμε γύρει αντιρρήσει όσον αφορά την προτινόμενη αυτή συγχώνευση, γιατί υπάρχει κίνδυνο μεγάλη συγκέντρωση ε, στην Αυστρία. Ελπίζω να διορθωθεί η κατάσταση και να μην ε, υπάρχει λόγος για ανησυχία στην περίπτωση αυτή τη συγχώνευσης για τις δημοσιονομικές υπηρεσίες τώρα. Και εδώ έχουμε αρχίσει δράσεις με έρευνες για καρτέλ όσον αφορά διάφορες δημοσιονομικές, ε, δημοσιονομικά ιδρύματα. Όπως για παράδειγμα για τον Ιαπωνικό δικτύο Τάιμπορ και όχι μόνο. Είναι πράγματα που έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτή την αίθουσα. Επίσης και όσον αφορά τα swaps, εξετάζουμε τι γίνεται σε διάφορες ε, τράπεζες, όπως επίσης και για τα CDS. Η δουλειά μας συνεχίζεται να ελέγχουμε δηλαδή τις κρατικές ενισχύσεις προς ε, τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δύο, την Ortel B και την Bayern B για παράδειγμα της Γερμανίας, την Ισπανική την UNIM από την TTUBA και το λουξεβοριακό τμήμα της Δέξια. Και βέβαια θα δούμε τι θα κάνουμε και για το υπόλοιπο τμήμα της Δέξια. Τώρα αναλύουμε επίσης τι γίνεται και με τον βελγικό κλάδο της Δέξια που είναι η Μπέλφιους. Και σε παραδοσιακούς κλάδους δραστηριοποιούμεθα και ασχολούμαστε με το τομέα του χάλιβα, συγχωνεύσει σε αυτό το τομέα, όπως επίσης και για την United Parcel Services, την UPS και την TT. Και ανάμεσα στην Glencore και την Extrata υπάρχει και εκεί κοινοποίηση. Στα ταχυδρομεία, η κρατική ενίσχυση έχει επίσης παίξει σημαντικό ρόλο Έχουμε πάρει πολλές αποφάσεις για την Deutsche Post, το B-Post, το La Post της Γαλλίας, τα ελληνικά ταχυδρομεία επίσης, τα βρετανικά. Και σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, το Deutsche Post, το γερμανικό και το, τη βελκική εταιρεία, μιλάμε για σύμβατη κρατική ενίσχυση. Ζητούμε πληροφορίες από τις εθνικές αρχές και έχουμε φτιάξει μια task force η οποία εξετάζει πιο πολλοί θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Μέσα στους επόμενους μήνες ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια συμπεράσματα από την Task Force προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις δράσεις μας τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Σε έναν άλλο τομέα τώρα, την φαρμακευτική βιομηχανία, η Λούμπε και η Σαρβιέ, δύο για δύο εταιρείε ε, γύραμε αντιρρήσει πριν από το καλοκαίρι, γιατί λέμε ότι κάνουν κατάχρηση ε, πατέντα στον τομέα των γενώσιμων φαρμάκων. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν οι πρακτικές αυτές σύντομα. Στις μεταφορές. Και εδώ ερευνούμε και μπορώ να σας πω ότι θα μας απασχολήσει πολύ αυτό ο τομέα στους επόμενους μήνες γιατί πρέπει να δούμε στον τομέα της ε, αεροπλοείας για παράδειγμα και να λύσουμε διάφορες περιπτώσεις που ήδη έχουμε ξεκινήσει να ερευνούμε. Υπάρχει και μια τρίτη προσπάθεια της ε, Ryanair να πάρει την Erlingus. Αυτή η συγχώνευση αναθεωρείται. Προσπαθούμε να βρούμε και λύσεις για προβλήματα που έχουν να κάνουν με συμμαχίε η SkyTeam και η START για παράδειγμα, με τον ίδιο τρόπο, Τέλο τέλος πάντων μια αντίστοιχη προσέγγιση όπως είχαμε κάνει παλιότερα. Τέλος, θα τελειώσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή όσον αφορά δράσεις για αποζημιώσεις από την νομοθεσία αντιτράστ. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να διευκρινίσει τη σχέση ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες παντού μέσα στην Ευρώπη να μπορούν να έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση λόγω βλάβης εξαιτίας παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από ότι εγώ πόσο δύσκολε είναι αυτέ οι συζητήσει, τόσο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσον αφορά τι συζητήσει που κάνουν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με του ε, συνομιλητέ μα είτε αυτοί είναι ε, ιδιωτικέ εταιρείε είτε είναι κυβερνήσει. Εσεί έχετε πει ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια πρωτοβουλία. Το είπατε και την τελευταία φορά στην έκθεση του Σάντζες Πρεσέδο. Συγχρόνως όμως γνωρίζετε πολύ καλά τι λέει και η έκθεση λένε που ψηφίσατε. Συνεχίζουμε λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συζητούμε τις εναλλακτικέ λύσεις που έχουμε. Σύντομα θα μπορέσω να έρθω και να σας παρουσιάσω περισσότερα πριν καταλήξουμε σε πρόταση που θα σταλεί και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε ερωτήσεις και θα απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις τώρα. Ακούτε τα ονόματα. Yeah. No. Uh, and I've got uh, Sophie. I've got Astrid as well. And I've got Dirk. Yes. Tremosa and Nicholas and yes, Bass. Anybody else? Πώς κανείς, Αλίσα. Αντολίν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Αντιπρόεδρο Αλμούνια για την παρουσία του και την παρέμβασή του έθεσε τρεις ε, στόχους. Ανάπτυξη, εξυγίανση των δημοσίων, οικονομικών και να συμβάλλει σε μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική αγορά. Είναι τρεις στόχοι τους οποίους εγώ συμμερίζομαι απόλυτα. Υπήρξαν δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι εν εξελίξη. Πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, προσφυγών επί τη βάση ζημιών λόγω βλάβης οικονομικής. Πρέπει εδώ να υπάρξει μια μεγαλύτερη διευκρίνηση της σχέσης του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα και μια απάντηση η οποία θα πρέπει να δοθεί για τις γενικευμένες αυτές ζημίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν στο θέμα των κρατικών επιδοτήσεων που είναι ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ε, ενεξελίξη μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ξέρω σε σχέση με τις ε, κατευθύνσεις που θέλει να ακολουθήσει η Κομισιόν για τις εταιρείε που βρίσκονται σε αναδιάρθρωση αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν, αν θα συμπεριλάβει και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες παραδείγματος χάρη, ή αν θα παραμείνουμε ειδική αντιμετώπιση και επίσης με ποιο τρόπο θα πρέπει να συνδεθεί αυτή η συζήτηση με τις συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα με ενδιαφέρει η δράση της Κομισιόν για τα επιτόκια αναφοράς. Αν θα μπορούσε λοιπόν να μας αναφέρει η Κομισιόν ποια είναι η γραμμή διερεύνησης που ακολουθεί, ποια είναι η γραμμή δράσης που προτίθεται να ακολουθήσει. Ξέρω ότι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει σημαντικές ε, παρεμβάσεις που αφορούν και τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα και την επίπτωσή τους στις απόρριές τους για την ε, ε, αγορά προϊόντων, για τα γενώσιμα προϊόντα, ακόμα και το software ανοιχτής πηγής. Θα ήθελα να ξέρω αν από τη δική του πλευρά ο κ. Σαρμούνια θα ήθελα να κάνει κάποια σχόλια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε επίσης και για, τις, ε, ε για τους κλάδους οι οποίοι έχουν χαρακτήρα δικτύου και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τροφιμικός τομέας, το τροφιμικό δίκτυο, γιατί φυσικά ένα πολύ σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού πηγαίνει σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να ξέρω αν έχει η Κομισιόν κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες επεξεργάζεται με τις ε, αρχές οι οποίες ασχολούνται με τα τροφιμικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Σαλμούνια. Αντολίν, να απαντήσω στις πέντε ερωτήσεις που μου έχει κάνει. Καταρχήν, οι προσφυγές λόγω ζημιών, για αποκατάσταση ζημιών κατά, καλύτερα, είναι μέσα στο πρόγραμμα της Κομισιόν. Ελπίζω ότι η πρωτοβουλία της Κομισιόν θα διατυπωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή που είναι γνωστή η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ε, ρύθμιση για την ε, ε, αποκατάσταση ζημιών σε μεμονωμένο επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας ζήτησε να νομοθετήσουμε για το θέμα αυτό για να μπορεί να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να καταμετρηθεί η έκταση της ζημίας και των πληροφοριών που μπορεί να έχει στα χέρια της Κομισιόν μια έρευνα παραγωγή σε καρτέλ που περιλαμβάνει και μέτρα επίοικειας για αυτούς που συνεργάζονται με τέτοιου είδους έρευνες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία και να την αποστείλουμε στο Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα είναι οι λεγόμενες συλλογικές προσφυγές. Υπάρχει μια έκθεση του Κοινοβουλίου, η έκθεση Μπελένε, η οποία μα έχει ζητήσει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό οριζόντια, όχι μόνο στα πλαίσια τη πολιτική ανταγωνισμού, αλλά σε όλε τι πτυχέ των συλλογικών προσφυγών. Φυσικά είναι διαφορετική κατάσταση σε ορισμένου χώρου από ό,τι σε άλλου σε ό,τι αφορά τι συλλογικέ προσφυγέ. Και υπάρχουν και κάποιοι τομεί που θεωρούν ότι δεν πρέπει να ρυθμίσει τα θέματα αυτά, να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ανοιχτή η συζήτηση και υπάρχει και η έκθεση του βουλευτή Σάντσεφ Πρεσέδο από την Οικονομική Επίτροπη που μας ζητάει την νομοθετική ρύθμιση σε όλες τις ε, πτυχές του θέματος και υπάρχει και μια άλλη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει εγκριθεί που ζητάει τα θέματα των συλλογικών προσφυγών να αντιμετωπιστούν με οριζόντιο τρόπο. Έχει λοιπόν ανοίξει και πάλι η συζήτηση Πιστεύω όμω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση και σίγουρα το Κοινοβούλιο ακόμα στην τρέχουσα θητεία θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει για τα θέματα αυτά και ελπίζω και να καταλήξει και σε νομοθετικέ ρυθμίσει. Τώρα, για την διάσωση επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωσή του. Εργαζόμαστε προ το παρόν για να αναπτύξουμε τι κατευθυντήρε γραμμέ για, για τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα όπου είναι απαραίτητο να επικαιροποιήσουμε τις κατευθύνσεις που ακολουθούμε μέχρι στιγμής. Για τον ίδιο τον πιστοτικό τομέα, <clears throat> τον τραπεζοπιστωτικό τομέα, πρέπει και εκεί να παρουσιάσουμε γενικές κατευθύνσεις, αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία μας επί τη βάση του πλαισίου που έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτό το διαχωρισμό. Θα προχωρήσουμε καταρχήν στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα και από τη στιγμή που θα είμαστε σε θέση να έχουμε στα χέρια μας ένα πλαίσιο το οποίο θα διέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε φυσιολογικές συγκυρίες, τότε θα είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε και τις κατευθυντήρες γραμμές για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Τι μένει τώρα εκρεμές σε αυτό το τομέα πέραν υποθέσεων που παραμένουν ανοιχτέ, όπως στην περίπτωση της Δέξια που μου είπατε βασικά είναι το θέμα της αναδιάρθρωσης με συμμετοχή του δημόσιου τομέα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως των τραπεζικών ε, συστημάτων χωρών όπως είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, που βρίσκονται μέσα σε κάποιο σύστημα μνημονίου ε, είναι πολύ πιθανό ότι και η Κύπρος θα προσταθεί στις τρεις αυτές χώρες γιατί ζήτησε ένα γενικό πρόγραμμα διάσωσης και στην Κύπρο φυσικά όπως ξέρετε το τραπεζικό σύστημα έχει ένα μεγάλο ειδικό βάρος στην οικονομία της και επίσης και σε ένα διαφορετικό επίπεδο εργαζόμαστε με την Ισπανία επί τη βάση του μνημονίου κατανόηση το οποίο ενεκρίθη αυτό το καλοκαίρι ώστε να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση μιας σειράς από χρηματοπιστωτικές οντότητες περίπου το ίμιση του τραπεζικού συστήματος της Ισπανίας θα συμπεριληφθεί σε αυτές τις ενέργειες. Προς το παρόν λοιπόν προχωρούμε σε μια ε, χωριστή αντιμετώπιση και είμαστε πιο προσεκτικοί εφόσον ακόμα δεν έχουμε καθορίσει το μελλοντικό οριστικό πλαίσιο για τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Για τα επιτόκια αναφορά, όπως σας είπα και πρόσφατα, έχουμε ξεκινήσει έρευνες σε σχέση με δυνατή ε, χρησιμοποίηση πρακτικών κάρτελ για τη χειραγώγηση της Libor, της Euribor και της Tibor. Είναι τρεις περιπτώσεις, αλλά δεν αποκλείω να υπάρξουν και περαιτέρω έρευνες. Αυτές οι ενέργειες είναι, κατά πέσα πιθανότητα, δράσεις οι οποίες έχουν χαρακτήρα καρτέλ, γιατί δεν είναι μονάχα χειραγώγηση, με πρόθεση χειραγώγηση, αλλά με πρόθεση να επωφεληθεί κανείς και από τη χειραγώγηση. Εργαζόμαστε επίσης πάρα πολύ για την βελτίωση των εργαλείων μας στον τομέα ανταγωνισμού, antitrust και επίσης στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων έχουμε τις ευραστεχνίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε πρότυπα τις ε, ευρεστεχνίες που περιλαμβάνονται λοιπόν σε συγκεκριμένα πρότυπα. Συνεργαζόμαστε με τις Αμερικανικές Αρχές Ανταγωνισμού και πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους και η αντιμετώπιση μας για αυτές τις περιπτώσεις όταν ο ιδιοκτήτης μιας ευρεστεχνίας που βρίσκεται σε ένα πρότυπο. Πότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάχρηση. Αυτό είναι το ερώτημα και εκεί έχουμε πιστεύω μια παράλληλη αντιμετώπιση ως Κομισιόν με τις Αμερικανικές Αρχές για τις ευρεσιτεχνίες εμπλέκονται επίσης και στον φαρμακευτικό τομέα, όπως είπαμε προηγουμένως. Είχαμε δύο περιπτώσεις για δύο εταιρείες και αυτά τα στοιχεία τα πρόκυψαν μετά από μία έρευνα που κάναμε το 2009. Στον φαρμακευτικό τομέα αφορά την Johnson και την Novartis μία περίπτωση και το άλλο ένα φάρμακο το οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιπτώσεις όπου προχωρούμε για θέματα ανταγωνισμού στο φαρμακευτικό τομέα και τέλος για τον τροφιμικό τομέα. Εγώ φυσικά έχω απόλυτη επίγνωση του ρόλου αυτό το τομέα για τον απλό πολίτη που κάθε μέρα θα πρέπει να πάει στην ε, αγορά τροφίμων και το καλάθι της νοικοκυρά σε μεγάλο βαθμό βαραίνει από τα τρόφιμα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, υπάρχουν προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Αλλά ακριβώ και για αυτό το ρόλο, λόγο, αυτό το οποίο οργανώσαμε, χάρη στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού, έχουμε οργανώσει μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε με τις ενέργειες που έχουν, κάνει, έχουν φέρει σε πέραση οι εθνικές αρχές, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη συνεκτικότητα μεταξύ των δράσεων των διαφόρων αρχών ανταγωνισμού και δεν είναι τυχαίο αυτό γιατί εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες που όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα και το αποτέλεσμα των ε, ε, εργασιών αυτής της ομάδας εργασίας μπορεί να μας δώσει και κατευθύνσεις για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο των αρχών ανταγωνισμού. και να ανοίξουμε και έρευνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σας λέω ότι μέχρι στιγμής είναι περιορισμένες αυτές οι έρευνες σε εθνική κλίμακα με ενιαίους κανόνες και έχουν και την, τα ίδια αποτελέσματα από ότι όταν του κάνει η Κομισιόν και όχι οι Εθνικές Αρχές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία που ξεκινήσατε ε, και για την Gazprom. Γιατί είναι ένα θέμα τεράστιας εμβέλειας. Και καλό θα ήταν να παρακολουθήσουμε τα τεκτενόμενα. Ενδιαφέρον είναι που άκουσα τις διάφορες προτεραιότητές σας. Σας παρακολούθησα με ευκολία και καταλαβαίνω τι θέλετε να κάνετε. Τα θέματα για των κρατικών ενισχύσεων, των καρτέλ και των αντιμονοπολίων. Πολλοί από τους κανόνες μας για τον ανταγωνισμό αφορούν το πώς θα οργανωθεί ο ανταγωνισμός και η επιχειρηματική ζωή που έχουμε. Όχι ο ανταγωνισμός και η επιχειρηματική ζωή που θα έχουμε στο μέλλον. Τι πιστεύετε κατά την άποψή ότι πρέπει να, να γίνει, ούτω ώστε εμείς και η Κομισιόν, ούτως ώστε να ελέγξουμε και να αναλύσουμε τα διάφορα, του διάφορους φραγμούς που έχουμε και στο εσωτερικό των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Κάποια από τα προβλήματα που αναφέρατε είναι λειτουργικά προβλήματα. Δηλαδή, σε ορισμένε χώρε είχαμε πολύ λίγο ανταγωνισμό. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα άκουγα από εσά να μου πείτε ποιε είναι, ποιες είναι κατά την άποψή σα οι ευκαιρίε που έχουμε για να αναλύσουμε πιο συστηματικό τρόπο τα, τους φραγμούς και αν τους ξεφορτωθούμε, ούτως ώστε να υπάρξει μια νέα κουλτούρα ανταγωνισμού και στο εσωτερικό των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Δεύτερο θέμα. Ναι, και είναι μεγάλο τμήμα της οικονομίας μας αυτό. Κάτι που είναι σημαντικό αλλά και πολιτικά ευαίσθητο. Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε τις τηλεπικοινωνίες ή τις, α, τους αερομεταφορείς ως ε, εταιρείε κοινή ωφελία, ας πούμε, γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Απαντώντας στον κ. Σάντζες ε, Πρεσέδο, μιλήσατε επίσης για τη σημασία του τομέα των τροφίμων. Αλλά αν συγκρίνουμε τώρα αυτόν τον τομέα με τις τηλεπικοινωνίες ή με τις αερομεταφορές, ε, τα τρόφιμα είναι ακόμα πιο σημαντικά για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Υπάρχουν ευκαιρίες για να εξασφαλίσουμε περισσότερο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί εδώ έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπου οι ευρωπαίοι πολίτες ε, εξαρτώνται από αυτές τις υπηρεσίες, από την αποτελεσματικότητά του, από τις υπηρεσίες που προσφέρονται και βεβαίω από το κόστος για τον νοικοκυριό. Τρίτον, κρατικές ανισχύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου στο χώρο αυτό. Ε, εξυγχρονίζοντας τις κρατικές ενισχύσεις, υπάρχουν και ευκαιρίες για να έχουμε λιγότερες αλλά πιο στοχευμένες ε, κρατικές ενισχύσεις. Λιγότερες, γιατί είναι σημαντικό για τους φορολογούμενους αλλά και για τις κυβερνήσεις που αγωνίζονται να περιορίσουν τα ελλείμματά τους. Είναι σημαντικό να είναι και πιο στοχευμένες ούτως ώστε και οι περιφέρειες και διάφορα τμήματα της Ευρώπης να επωφεληθούν όχι μόνο από περισσότερο ανταγωνισμό, αλλά να αναπτυχθούν ε, και εκεί όπου υπάρχουν μειονεκτήματα, δηλαδή εκεί που έχουμε μειονεκτούσες περιοχές, να αναπτυχθούν χάρη στον ανταγωνισμό. Μάλιστα, η φραγμή στην είσοδο είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, το, ο πιο σημαντικός φραγμός που θα ήθελα να φύγει όταν μιλάμε για τις ε, περιπτώσεις αντιτράστ στο εσωτερικό των κρατών μελών. Σε ορισμένε περιπτώσει αντιμετωπίσαμε τέτοια θέματα ε, στο πρόσφατο παρελθόν. Παραδείγματο χάρη με τις τηλεπικοινωνίε. Και μας ε, υποστήριξε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με μία απόφαση. Ε, σε μία περίπτωση εναντίον της τηλεφώνικα, της ισπανικής ε, τηλεφώνικας, γιατί πίεσε την αγορά και προσπάθησε να μην ε, αφήσει άλλους ανταγωνιστές να μπουν στην αγορά ή να τους δημιουργήσει δύσκολες ε, συνθήκες. Αυτά ήταν για την Ισπανία. Είχαμε και άλλες ε, περιπτώσεις με τέτοια προβλήματα μεταξύ κρατών μελών, όχι στο εσωτερικό κρατών μελών πια. Η Gazprom, Φερρυπίν, στην οποία αναφερθήκατε. Η πρώτη ανησυχία που είχαμε όταν ξεκινήσαμε την έρευνα για τις δραστηριότητες της Gazprom στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ήταν η δυνατότητα να επιβάλλουν κατά κερασμό της αγοράς του αερίου, γιατί υπάρχουν διάφορες ρήτρε με τους αγοραστές εδώ στα κράτη-μέλη προσπαθώντας να δημιουργήσουν εμπόδια και να μην ε, επιτρέψουν την επανεξαγωγή του αερίου από την Πολωνία, ας πούμε, που αγοράζεται από την Πολωνία, από την Τσεχία κτλ. Ή σε άλλες χώρες. Και τα εσωτερικά εμπόδια ή και τα συνοριακά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ενή αγορά και τα αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζουμε τέτοιου ε, εμπόδια σε πολλέ από τις υποθέσεις που ερευνούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Υπηρεσίε Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Δεν μιλάω μόνο για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε δίκτυο. Όπως ξέρετε, πέρυσι υιοθετήσαμε το νέο πλαίσιο ή μήπως ήταν στις αρχές του 2012. Δεν θυμάμαι αν ήταν ε, Δεκέμβριος του 2011 ή Ιανουάριος του 2012. Υιοθετήσαμε λοιπόν το νέο πλαίσιο για τις ε, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος για να αξιολογήσουμε το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, συμβατότητα των δημοσίων επιδοτήσεων για τη χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων και την προστασία των κανόνων του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς. Και είπαμε ότι θα πρέπει να συνδέσουμε αυτές τις α, υπηρεσίες με το επίπεδο α, πληρωμής αυτών των υπηρεσιών. Αυξήσαμε το κατόφλι κάτω από το οποίο δεν πληρώνουμε, ας πούμε, δεν, δεν δίνουμε σημασία, γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχει σημασία για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για τις διασυνοριακές σχέσεις. Από την άλλη, οι μεγάλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν έχουν να κάνουν με τον αρχικό υπολογισμό της αποζημίωσης, της πληρωμής, εν σε αντιδιαστολή με την επιδότηση και το κέρδος, αλλά πρέπει να δούμε και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών. Μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό. Και σε περίπτωση που έχουμε ωφέλη, λόγω αποτελεσματικότητας, ποιος επωφελείται, ο πάροχος ή ο πολίτης. Νομίζουμε ότι φτιάξαμε μια σωστή εξίσωση εδώ. Μια καλή ισορροπία πετύχαμε. Μιλήσατε για τις αεροπορικές εταιρείες και τον τομέα των αερομεταφορών. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές. Είναι και πολύ σημαντική συζήτηση, αλλά και δύσκολη αυτή. Από τη μία, μιλάμε για επιδοτήσεις για νέες επενδύσεις, αλλά και για λειτουργικά έξοδα, για τα τοπικά και περιφερειακά αεροδρόμια. Και πρέπει να αποφασίσουμε πότε και υπό ποιους όρους η ενίσχυση για επενδύσεις σε νέα αεροδρόμια συνάδει με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Και μήπως αυτές οι επενδύσεις αν βελτιώνουν την διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση ας πούμε, των εδαφών μας και των περιοχών μας ή μήπως αυτές οι κρατικές ενισχύσεις για τα περιφερειακά αεροδρόμια μπορούν να δημιουργούσουν αθέμητο ανταγωνισμό ε, με ήδη υπάρχοντα αεροδρόμια. Ε, συνήθως αυτά τα τοπικά περιφερειακά αεροδρόμια ε, συνδέονται με εταιρείες χαμηλού κόστους. Έτσι, εκεί πετάνε κυρίως αυτές οι εταιρείες. Αυτή είναι πολύ σημαντική συζήτηση. Από την άλλη έχουμε και τις κλασικές αερο εταιρείε αεροπονικών μεταφορών που έχουν πάρα πολλέ δυσκολίε αυτή την εποχή. Θα πρέπει να έχουμε ε, μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτέ τι ε, εταιρείε χαμηλού κόστου που επιτρέπουν σε εκατομμύρια επιβατών Ευρωπαίων να πετάξουν, αλλά από την άλλη να έχουμε σωστό ανταγωνισμό ανάμεσα στι κλασικέ μεταφορικέ εταιρείε και στι εταιρείε χαμηλού κόστου. Επίση, λιγότερε κρατικέ ενισχύσει, αλλά πιο στοχευμένε. Ναι, το συζητάμε. Και στο νέο πλαίσιο που συζητάμε όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, περιφερειακή ενίσχυση για να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ευρώπη. Αυτή τη βδομάδα όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι εδώ στις Βρυξέλλες. Για αυτή την ημερίδα με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουμε. Και συζητάμε τις ε, νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις, περιφε... τις ε, περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις. Μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Επίτροπο Χάν, θα συζητήσουμε αυτές τις περιφερειακές ενισχύσεις. Πρέπει όλες τις ενισχύσεις αυτές να τις βάλουμε σε ένα καλάθι. Όχι. Πρέπει να προστατεύσουμε τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες ενισχύσεις για να προσελκύσουν επενδύσεις και να εξασφαλίσουμε και μια μεγαλύτερη ισοτιμία και να μην επιτρέπουμε πάντα τις καλές επενδύσεις να τις καρπώνονται, ας πούμε, οι πιο πλούσιες ε, περιφέρειες. Προφανώς. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες, να δούμε πού δεν λειτουργεί η αγορά, να την καταλάβουμε καλύτερα και να δούμε πού παίζει ρόλο στο που συσσωρεύονται οι επενδύσεις. Επίσης, ποιο είναι το κατάλληλο ύψος έντασης επένδυσης που θεωρείται συμβατό πώς μπορούμε να μοιράσουμε αυτή την ένταση των επενδύσεων, δηλαδή σε περιφέρειες που είναι κάτω από το 75% του κοινοτικού ΑΕΠ ε, κατά κεφαλή και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, περιφέρειες που είναι πάνω από το 75% αλλά κάτω από το κοινοτικό μεσόωρο. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα θέματα, πολύ δύσκολε συζητήσεις και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από τη μία τις δυσκολίες των εθνικών προπολογισμών και των περιφερειακών προπολογισμών. Άρα πρέπει να είμαστε πιο ακριβεί και ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι σε μια περίοδο κρίση όλοι όσοι μπορούν να προσελκύσουν επενδύσει θα έχουν περισσότερε ευκαιρίε για να ξεπεράσουν τι συνέπειε τη κρίση. Και επομένω. Αυτή πάντα είναι δύσκολη συζήτηση, αλλά σε περίοδο κρίσης γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Και ελπίζω να το καταλάβετε αυτό βλέποντας και την τελική απόφαση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σόφη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε πάλι εδώ και έχουμε αυτή την καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Θα είμαι σύντομη. Για τις κρατικές ενισχύσεις. Αναφερθήκατε στο ότι σκέφτεστε να ευρύνετε τις εξαιρέσει στον κανονισμό. Αλλά θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει στην Επιτροπή μας εδώ, που είχατε πει ότι η έκθεση δείχνει πως 40%, 40% των περιπτώσεων ε, βάζουν ερωτηματικά κατά πόσο αιτιολογούνται δηλαδή ή όχι. Ε, αυτό δεν θα έπρεπε να το δούμε πιο πριν, πριν βρίνουμε το πεδίο εφαρμογή των εξαιρέσεων αυτών. Δεύτερον, πώς υπαλληφεύεται την επίδοση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στα πλαίσια αυτού του δικτύου που λέγατε. Άκουσα τον Χούκαν Χόκμερ για τις μεγάλες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα είδα για την Ολλανδία, για μια επιχείρηση φέρει που με τη στήριξη των αρχών ανταγωνισμού κάνει προσπάθειες να εμποδίσει την είσοδο νέων στην αγορά. Ε, λοιπόν, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. Εσείς πώς το παληθεύετε αυτό. Γιατί το σύστημα είναι τόσο δυνατό όσο πιο δυναμός κρίκος. Άλλα θέματα τώρα, αντιτράστ και καρτέλ. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της Google. Πρέπει να σας πω ότι εμεί πολλές φορές τα θέτουμε και ζητάμε να γίνονται ανατομέα έρευνες. Είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς για ποιο τομέα μιλάμε, γιατί είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι εντελώς νέες και μοναδικές. Τα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, κοινωνική δικτύωση. Το Facebook αυτή τη βδομάδα είπε ότι έχει ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Ένα δισεκατομμύριο, δηλαδή ένα στους στον ε, τομέα αυτό, στον ε, κόσμο αυτό, χρησιμοποιεί το Facebook. Ε, δεν είναι τελικά μονοπόλιο, δεν υπάρχουν πραγματικοί ανταγωνιστές και έχουν και τεράστια δύναμη. Άρα, οπότε αναρωτιέμαι, μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ανησυχίες. Δηλαδή με, με ανησυχεί το γεγονός αυτό ότι υπάρχει μια εταιρεία που έχει ένα δισεκατομμύριο χρήστες, άρα τεράστια δύναμη πώς να εφαρμόσουμε τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την επιλογή του καταναλωτή κτλ. Αναρωτιέμαι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σκέφτεται καθόλου πώς να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες μορφές μη παραδοσιακές που έχουμε μπροστά μας, αυτούς τους νέους τομείς. Έχω την αίσθηση ότι εξακολουθούμε να τους βλέπουμε αυτούς τους νέους τομούς σαν ε, κάποιες προσπάθειες startup ε, εταιρείε που κάνουν ε, φοιτητέ και έτσι νέοι. Δεν λέω ότι θέλω να τους κόψουμε τα φτερά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε στα σοβαρά που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Και νομίζω ότι μιλάω ε, μέρους όλων. Και, και διακόπτω δε πρόεδρος, ναι, ναι, το καταλάβανα ότι είχατε άλλη μια ερώτηση, αλλά να είναι και τελευταία σας. Ναι, λέει η κυρία Φαντερβέλτ. το θέμα των ε, καρτών πληρωμής. κάτι για παράδειγμα. Πάντα λέμε ότι αργεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά θα είναι αδύνατον να υπάρχει είσοδος νέων ε, στην αγορά και να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός και εδώ. Ο Επίτροπος, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, σύντομα, να μην εδώ πέρα έχω την πρόεδρο να με προειδοποιεί με το σφυράκι της. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι συμβατό από τη μια μεριά να έχουμε τις γενικές εξαιρέσεις και να καλύπτουμε τους τομείς εκείνους που θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε κοινοποίηση για την ενίσχυση, γιατί θεωρούμε, εκτός αν υπάρξει βέβαια κάποια προσφυγή, θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ε, στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προγράμματα. Συγχρόνως, μπορούμε να είμαστε πιο αυστηροί από ό,τι είμαστε τώρα ε, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι φέρνουν σε πέρα τις υποχρώσεις τους. Γιατί αυτό είναι δικιά μας αποκλειστική ευθύνη. Αλλά πρέπει να σέβονται τους κανόνες, να ελέγχουν οι εθνικές αρχές δηλαδή τα διάφορα προγράμματα και να επιβεβαιώνουν ότι δεν αντιβαίνουν τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και να φροντίσουν να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, πολλές χώρες μέλη το κάνουν και μάλιστα οργανώνουν τις διαδικασίες τους και τις αποφάσεις που παίρνουν, τις παίρνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο έγκυρα είναι τα διάφορα προγράμματα και συνάδουν με τους κανόνες για τις κρατικές επιχειρήσεις, ενισχύσεις. Άλλες χώρες δεν το κάνουν τόσο. Έχετε δίκιο ότι από την πρώτη ανάλυση για το τι γίνεται με τα προγράμματα που δεν υπόκεινται σε κοινοποίηση, όντω υπήρχε αυτό το 40% που είδαμε ότι δεν συμμορφώνεται. Και συγχρόνω η ενίσχυση για φυσικέ καταστροφές ή για δασοκομεία ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κάτι καλό για την καλή ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προσπαθούμε πάντως να επικεντρωνόμαστε καλύτερα σε ό,τι είναι πραγματική προτεραιότητα. Και πιστεύω ότι είναι συμβατά αυτά τα δύο μεταξύ τους. Γι' αυτό και προσπαθούμε να καλύψουμε και τις δύο πλευρές. Λιγότερη παρέμβαση από την πλευρά μας, δηλαδή όταν έχουμε μικρές περιπτώσεις. Και περισσότερη προσοχή στο με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη φέρουν σε πέρα στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των ε, κρατικών ενισχύσεων. Τώρα, πώς να επαληθεύσουμε την ποιότητα μιας εθνικής αρχής ανταγωνισμού. Μα υπάρχει το δίκτυο αυτό που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και λειτουργεί και πάρα πολύ καλά. Η εμπειρία μας είναι πολύ θετική. Αυτός ο συντονισμός που γίνεται Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Αρχών πρέπει να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες, αυτούς που έχουμε από τη συνθήκη και η εμπειρία μας στο συντονισμό αυτό είναι πολύ θετική. Βέβαια, αν η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού υιοθετήσει αποφάσεις και εφαρμόζει το 1 ή το 1-2 της συνθήκης, εμείς δεν μπορούμε να διορθώσουμε τις αποφάσεις τους, πρέπει να τους πάμε στο δικαστήριο, κάποιος είτε στα εθνικά είτε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Πάντως, το δίκτυο αυτό ευρωπαϊκού ανταγωνισμού με ικανοποιεί ως προς τον τρόπο που λειτουργεί. Κοινωνική δικτύωση τώρα. Όπως είπα και πριν απατώντας σε κάποια άλλη ερώτησή σας μια άλλη φορά, η Google είναι ένας τομέας από μόνος του. Αυτό που κάνουμε με το Google είναι μια έρευνα που κάνουμε για τον τομέα αυτόν, γιατί είναι μια νέα δραστηριότητα. Κοινωνικά δίκτυα επίσης είναι ένας ε, τομέας με τεράστια δυναμική και δυναμισμό. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, δεν ξέρω. Στο μέλλον, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί. Αλλά δεν ξέρω τι δίκτυα τέτοια θα προκύψουν για να δούμε κατά πόσο τηρούν τους κανόνες τους αντιμονοπολιακούς ή όχι. Προς το παρόν παρακολουθούμε και όχι μόνο το θέμα των μονιπολίων, αλλά και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό βίο, με την προστασία του καταναλωτή επίσης. Είναι όμως ένας πολύ δυναμικός τομέας που προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε, ακόμα και αν δεν έχουμε ε, τέτοια υπόθεση υπό έλεγχο. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία προσφυγή, κανένα παράπονο, δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα κοινωνικού δικτύου που να ελέγχουμε, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα υπάρξει μια τέτοια υπόθεση να ελέγξουμε. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και δεν είναι μόνο θέμα ψυχαγωγίας για το πώς θα επικοινωνούμε με τους φίλους μας και οικονομικά είναι ένας τεράστιος τομέας. Διακυδεύεται πάρα πολύ χρήμα. Οι πληρωμές τώρα και οι κάρτες ε, πληρωμής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας επιβεβαίωσε τη θέση μας όσον αφορά την υπόθεση Mastercard. Έχουμε και παραπάνω στοιχεία για την Visa Europe πάντα ο Μισελ Μπαρνιέ και εγώ ίδιος από κοινού ξεκινούμε διαβούλευση για τη νέα γενιά πληρωμών, συστημάτων πληρωμών με κινητά, με κάρτες κλπ. Και τις προάλλες συναντήθηκα μαζί του και με τις υπηρεσίες μας για την παρακολούθηση του θέματος. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, στην περίπτωση των καρτών, των πιστοτικών και των πληρωμών, ε, αλλάζουν πολύ συχνά τα τέλη, όπως και στη Βίζα. Και η καλύτερη λύση, κατά πάσα πιθανότητα, είναι η ρύθμιση. Αυτό συζητούσαμε το Μισελ της προάλλες. Δεν ξέρω πότε, αλλά σίγουρα θα προχωρήσουμε σε κάποια σχετική πρωτοβουλία. Ωραία. Θα είμαι σύντομος, ο Μπάρτ λέει. Μην τρομάζετε. Τρία ερωτήματα έχω να θέσω. Πρώτα απ' όλα, για την τέξια. Αναφερθήκατε στην τέξια και είπατε ότι θα υπάρξουν και κάποια άλλα πακέτα διάσωσης για τις κυπριακές και ισπανικές ε, τράπεζες που επίκυνται. Το ερώτημα μου είναι, όταν έγινε σαφές ότι η πρώτη αναδιάρθρωση στην τέξια δεν ήταν επιτυχής, τι μπορούμε να αποκομίσουμε ως εμπειρία. Φαντάζομαι ότι εσείς στην Κομισιόν έχετε προχωρήσει σε μια ανάλυση, μια εσωτερική αξιολόγηση του τι πήγε στραβά και ίσως μπορούμε να επωφεληθούμε όταν πρέπει να κάνουμε αναθιαρθρώσεις άλλων τραπεζών. Αν έχετε να μας πείτε λοιπόν ποια διδάγματα έχετε αποκομίσει από την πρώτη αναδιάρθρωση της Δέξια. Δεύτερον, για την, τον εξυγχρονισμό των κρατικών επιδοτήσεων. Μιλήσατε για τις προδιαγραφές για το περιβάλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είπατε ότι αυτή η επικαιροποίηση θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους της ε, Ευρώπης 2020, όπως είναι κλιματική στόχοι, στόχοι ενέργειας. <clears throat> Πώς θα εμφανιστούν λοιπόν αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές για να υποστηρίξουν την ανανεώσιμη ενέργεια και την ε, ενεργειακή ε, αποδοτικότητα. Τρίτον, αναφέρθηκε το θέμα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Και αυτό φυσικά είναι ένα ειδικό θέμα για τις κάτω χώρες, αλλά ξέρω ότι και στη Γαλλία υπάρχουν προβλήματα με την κοινωνική στέγαση. Ξέρουμε ότι όταν πρόκειται για εξαιρέσει. Υπάρχει και εδώ κάποιο περιθώριο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από τους κανόνες κρατικών επιδοτήσεων. Βλέπουμε τώρα στις κάτω χώρες, και το γνωρίζετε αυτό φυσικά, γιατί αναφέρθηκε και στο παρελθόν, για πολλές για πολλά νοικοκυριά δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα λόγω των κανόνων της Ολλανδικής Κυβέρνησης και της Κομισιόν. Μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πάρετε μια ευέλικτη και επικοδομητική στάση έναντι κρατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κοινωνική στέγαση λόγω της υπερβολικά στενής ερμηνείας που γίνεται. Αν σας ζητήσει λοιπόν η Ολλανδική κυβέρνηση μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι ήμουν σύντομο. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Αλλά η περίπτωση της δέξια δεν μπορεί να καλυφθεί σε ένα λεπτό. Τι πήγε στραβά. Το πρόβλημα με τη δέξια τηλεγραφικά είναι ότι ήταν υπερβολικά πολυδάπανη η χρηματοδότησή τους και προσπαθούσαν συγχρόνως να παρέχουν φτηνή πίστοση. Κόστιζε πάρα πολύ η χρηματοδότησή της, ενώ οι δανειοδοτήσει τη δεν ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρε. Επομένω, δεν ήταν βιώσιμη η λειτουργία αυτής τη επιχείρησης. Τι κάνουμε εμεί. Υπάρχει το σχέδιο περαιτέρω αναδιάθρωση, το πρώτο σχέδιο μάλλον αναδιάθρωση το 2010. Δεν εφαρμόστηκε σωστά, οι συνθήκε στην αγορά δεν ήταν τόσο ευνοϊκές όσο είχε θεωρηθεί ότι θα είναι όταν ελήφθησαν οι αρμόδιες αποφάσεις. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε σε δεύτερο γύρο την περίπτωση της Δέξια. Η, πολίθηκε η BIL στη, στο Λουξεμβούργο. Η Belfius, ο βελγικός κλάδος της Δέξια, έχει εθνικοποιηθεί πλήρως από την βελγική κυβέρνηση και περνάει μια αναδιάρθρωση. Και αυτό το οποίο μένει είναι η Δέξια Credit Local που έχει τα στοιχεία ενεργητικού από το παρελθόν. Και συζητάμε τη μία πλευρά από τη Βελική κυβέρνηση το πώς θα γίνει η αναδιάθρωση της Μπέλφιους και επίσης με τη βελική και γαλλική κυβέρνηση το πώς θα γίνει η αναδιάθρωση και η επίλυση σε κάποιο βαθμό του υπολείπου της, του ομίλου Δέξια με την Δέξια Κρεντή Λοκάλ. Έχουμε προχωρήσει σημαντικά στον τομέα αυτό. Δεν έχουμε τελειώσει βέβαια τις διαπραγματεύσεις όπως σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να περατώσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις γιατί δεν έχουμε ακόμα τις προτάσεις που χρειαζόμαστε και αυτές οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν σε εμά από τους ιδιοκτήτες του ομίλου Δέξια, τα κρατημέλη δηλαδή τη Γαλλία και το Βέλγιο, που έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν σημαντικές ε, Δυσκολίε στις συζητήσεις τους για το πώς πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ τους οι κρατικές εγγυήσεις που υποστηρίζουν τα υπολείμματα του ομίλου Ντέξια. Είναι πολύπλοκη συζήτηση, ελπίζω ότι είμαστε κοντά στο τέλος αυτής της διαδικασίας που θα μας οδηγήσει σε νέες αποφάσεις για τα διάφορα τμήματα του ομίλου Ντέξια. Αλλά όλα αυτά δεν περνάνε μόνο από το χέρι της Κομισιόν εξαρτώνται κυρίως από τους ε, ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των διαφόρων τμήματων που απαρτίζουν τον ομιλοντέξια. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε την ε, ε, απάντησή μας, αλλά αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει τι δικέ του προτάσει. Δεν μπορούμε εμεί να προτείνουμε λύσει. Πρέπει οι ιδιοκτήτε να το κάνουν αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Δεν έλεγα ειδικά για την δέξια. Τι μάθαμε από τα λάθη που έγιναν με την τέξια όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλε τράπεζε μέσα στην Κομισιόν τα λάθη. Η γενική μου εντύπωση ότι τα κάναμε θαυμάσια, ότι ήταν πολύ σωστή η αντιμετώπιση μα. Δεν έχουμε την αρμοδιότητα για επίλυση τραπεζών. Τα συζητάτε τώρα. Την πρόταση, επί τη βάση της ε, πρότασης λοιπόν της Κομισιόν, σε μια μελλοντική τραπεζική ε, ένωση, να προχωρήσουμε και περισσότερο για να έχουμε και αρμοδιότητα, δικαιοδοσία επίλυση. Εφόσον δεν έχουμε αυτή την δικαιοδοσία, τον Οκτώβριο του 2008 αναγκαστικά να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό μηχανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε τότε μετά την χρεοκοπία της Lehman Brothers για να έχουμε τις αρχές οι οποίες είχαν άλλο χαρακτήρα να λειτουργήσουν σαν αρχές επίλυσης. Αλλά στην δέξια. Αν δεν έχουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις αυτών που είναι υπεύθυνοι, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για λογαριασμό τους. Ακόμα και με αυτές τις πολύ σοβαρές δυσκολίες που έχουμε, παρόλα αυτά καταφέραμε να εγκρίνουμε αποφάσεις για τα σχέδια αναδιάρθρωσης περίπου 50 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συστάμε τώρα την πλήρη αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο την αναδιάρθρωση του μεγαλύτερου μέρους του πορτογαλικού συστήματος, τραπεζικού συστήματος, όλου του Ιρλανδικού συστήματος, του μισού συστήματος του Ισπανικού και αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κυπριακό σύστημα και ίσως και ένα τμήμα του σλοβενικού τραπεζικού συστήματος. Πέραν αυτό όμως έχουμε εγκρίνει αποφάσεις για τον τομέα των Landesbank και στη Γερμανία που είχε προβλήματα εδώ και πολύ καιρό και έχουν ε, περάσει τη διαδικασία αναδιάθρωσης, εν μέρη με επίλυση. Επίσης, αναδιαθρώσεις στον τραπεζικό τομέα για ορισμένε τράπεζες της Αυστρίας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το έργο που έχουν φέρει σε πέρας οι αρχές της Κομισιόν με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έπρεπε να πληρώσουν ακόμα περισσότερο ως φορολογούμενοι για την αναδιάθρωση του τραπεζικού τομέα για το περιβάλλον και τις κατευθυντήριες γραμμές. Μακρυγόρισα στο πρώτο ερώτημα, δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ίσως στην επόμενη συζήτηση που θα έχουμε μαζί, μας, μαζί σας, ίσως έχω να σας πω λίγο περισσότερο. Είμαστε απλώς στο σημείο εκκίνησης. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς θα αποφασίσουμε για τις ανανεώσιμες ενέργειες και αυτό που έχουμε προβλέψει είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις επιδοτήσεις σε βιομηχανικούς κλάδους που έχουν ένταση εργασίας που θα πρέπει να αποζημιωθούν για την αλλαγή στο σύστημα εμπορίας εκπομπών που θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο χρόνο. Λένε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν τη λεγόμενη διαρροή άνθρακος, δηλαδή την εγκατάσταση επιχειρήσεων. Κανείς δεν μου έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένα τέτοιο ε, πρόβλημα, αλλά εμεί έχουμε εγκρίνει κατευθυντήρες γραμμές που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα επακριβεί και αυστηρέ με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν τι προποθέσει κάτω από τι οποίε ορισμένε βιομηχανίε επειδή πρέπει να πληρώσουν μεγαλύτερο τίμημα ενέργεια λόγω του νέου συστήματο ETS, εμπορίας εκπομπών δηλαδή, μπορούν να τύχουν αποζημίωση από τι αρμόδιε αρχές. Και κοινωνική στέγαση μονάχα δύο λόγια να πω. Στο νέο πλαίσιο που έχουμε διατυπώσει, τονίσαμε ότι δεν είναι μια κοινοποιήσιμη υπηρεσία γενικού συμφέροντος η στέγαση. Υπήρξε μια περίφημη υπόδοση στην, ε, ε, στις κάτω χώρες λόγω ε, που διατυπώθηκαν την εποχή που ήταν αρμόδιος ο προκάτοχός μου ή προκατοχός μου. Τώρα η νέα κυβέρνηση στις κάτω όταν σχηματιστεί, δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη, θέλαν από μένα να παίξω το ρόλο του Υπουργού Στέγασης των Κάτω Χωρών. Είπα όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτή η δουλειά και δεν είμαι υποψήφιο. Δικό σας παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ας επιστρέψουμε στη χώρα σας, ε, κύριε Επίτροπε. Αναφέρατε τις ε, κρατικές ενισχύσεις και τον τομέα των τραπεζών. Πάω στην Πάνκια. Μια μικρή ερώτηση. Ποια ήταν η δική σας συμμετοχή, η εμπλοκή ως Επίτροπος Ανταγωνισμού στη δημιουργία της Μπάνκια, που είναι συγχώνευση 7 περιφερειακών τραπεζών, όπως ξέρετε. Σχολιάσατε, εγκρίνατε την ε, δημιουργία της Μπάνκια. Και αν ναι, τι ακριβώς κάνατε, ε, ακριβώς, επακριβώς. Απλή απάντηση. Δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν είναι πλάκιν καθόλου σε αυτή την υπόθεση. Ο Νικόλας είναι εδώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αλμούνια, συζητήσαμε για τις κρατικές ενισχύσεις. Επίσης, κάνετε νήξεις για χώρες που συναντούν δυσκολία, με έναν εφημισμό, εν πάση περιπτώσει. Να σας πω λοιπόν ένα δραματικό γεγονός επίκαιρο, αλλάζοντας αυτά που ήθελα να σας ρωτήσω και θα ήθελα να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Αναφέρομαι στους εργαζόμενους τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τα ναυπηγεία αυτά στο παρελθόν είχαν πάρει κρατικές ενισχύσεις. Λόγω των κρατικών ενισχύσεων η Κομισιόν απαγόρευσε στα ναυπηγεία να ναυπηγούν εμπορικά πλοία και πολεμικά πλοία εκτός από τα πολεμικά πλοία του πολεμικού ελληνικού ναυτικού. Τέτοιες παραγγελίες σήμερα δεν υπάρχουν. Τα ναυπηγεία είναι σε αδίέξοδο. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα και είναι απλήρωτοι για μήνες. Προχτές, λόγω της οργής, μπήκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα διαδηλώνω. Σας έχω ρωτήσει για αυτό το γεγονός και μου έχετε απαντήσει ότι λυπάσαστε για αυτές τις εξελίξεις, αλλά αν δεν υπάρξει επιστροφή από την Ελλάδα των παράνομων ενισχύσεων, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα ως προς αυτό. Στο μεταξύ υπάρχει μεγάλη ανεργία και μεγάλος τιμός. Εδώ είστε ο Επίτροπος Αλμούνια αλλά είστε και Ισπανός πολιτικός και δεν μπορώ να σας μιλήσω παραπάνω για την ανεργία που η χώρα σας είναι πρωταγωνίστρια και για την αγανάκτηση που έχει ο κόσμος στην Ισπανία. Και σας ερωτώ, είναι δυνατόν να μένετε στη δικαιολογία ότι η Ελλάδα δεν έχει επιστρέψει τις ενισχύσεις Τυπικά έχετε δίκιο. Τυπικά έχετε δίκιο. Αυτή είναι η νόμη. Αλλά είναι νόμη να μου επιτρέψετε του ισχυρού που μα οδηγούν στην κοινωνική ζούγκλα. Αυτή είναι η νόμη. Περιμένετε από την Ελλάδα σε αυτή την οικονομική κατάσταση που σα είναι γνωστή να του επιστρέψει. Θα μείνετε σε αυτό το σημείο. Σα ερωτώ λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή. Υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω, έχετε και μια συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξη τη Ελλάδα νομίζω αύριο. Υπάρχει περίπτωση να εξετάσετε την περίπτωση να αρθεί αυτή η απαγόρευση, ούτω ώστε να υπάρξει δουλειά σε αυτή την, στον τομέα για να μπορέσουμε να φύγουμε από τα δραματικά αδιέξοδα που προσπάθησα όσο γίνεται πιο σύντομα να σας περιγράψω και που σας είναι γνωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, been uh, with this case the... Ασχολήθηκα σε διάφορες φάσεις με αυτή την υπόθεση. Είναι μια απόφαση μια απόφαση υιοθετήθηκε, αν θυμάμαι καλά, ούτω ώστε να μπορέσουν αυτά τα ναυπηγεία να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κατασκευής ε, αμυντικών πλοίων του πολεμικού ναυτικού, αλλά όχι του εμπορικού ναυτικού. Αυτή ήταν η απόφαση. Και στη δική μου χώρα, στην Ισπανία, ελήφθη παρόμοια απόφαση δεν είναι η μοναδική απόφαση προ αυτήν την κατεύθυνση που ελήφθη αυτή. Και μία απόφαση όταν λαμβάνεται θα πρέπει να εφαρμόζεται. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά δεν μπορώ να επιλύσω αυτές τις δυσκολίες λέγοντας δημόσια ότι δεν με ενδιαφέρει να εφαρμοστεί η απόφαση για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την Ελλάδα και σε άλλε χώρε δεν μπορούν να λυθούν με αυτόν τον τρόπο. Έχω τρει ομιλητέ στον κατάλογο. Άστριντ, Ελίζα και Ραμόν. Άστριντ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και εγώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για την τέξια, μια και μιλήσατε για αυτό το θέμα. Ακούσαμε το καλό νέο ότι η Δέξια που πέρασε σε φάση εξυγίανσης από το 2011 ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι η λουξεμβουργέζικη θηγατρική κατά 90% εφ' θα ανήκει στον εμμύρη του Κατάρ και κατά 10% στην ε, κυβέρνηση του Λουξεμβούργου. Έχουμε τα 730 εκατομμύρια που πλήρωσαν ε, από το Κατάρ. Αλλά εσείς συμφωνήσατε με αυτήν την απόφαση. Δεν ε, θεωρήσατε ότι η τιμή αυτή ήταν εξευτελιστική για να αγοραστεί αυτό το μερίδιο της Δέξια. Έχω και άλλα προβλήματα όμως γιατί το γαλλικό και βελγικό τμήμα της Δέξια χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση. Και το πρώτο εξάμεινο του 2011 έχασαν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπατε ότι δεν ξέρετε τι θέλουν να κάνουν, αλλά στις 27 Σεπτεμβρίου επιτρέψατε την παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2003 13 της προσωρινής εγγύησης των 55 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε δώσει ε, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και το Βέλγιο, ούτω ώστε να επιτρέψουν την ε, διάλυση του ομίλου. Μια και το Λουξεμβουργέζικο τμήμα έχει πολιθεί, η Λουξεμβουργέζικη κυβέρνηση θα πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσει να συμμετέχει στην εγγύηση το 55 αυτών δις. Κατά 3% η, συμμετοχή του Λουξεμβούργου είναι 3% στα 55 δις δηλαδή. Αν το Βέλγιο και η Γαλλία δεν μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους, τότε ο κύριος Γιούνκερ θα χρεοκοπήσει. Αν πρέπει να πληρώσει με βάση τον προϋπολογισμό του κράτους, ο οποίος είναι ήδη ελληματικός Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα που ακούστηκε. Το, ο τρόπος με την οποία η Eurostat αντιμετωπίζει το ποσοστό που θα πρέπει να πληρώσει η Γαλλία και το Βέλγιο σε αυτή την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης. Αν η Eurostat θεωρεί ότι η παρέμβαση είναι δαπάνη κρατική, τότε το Βέλγιο, η Γαλλία και ενδεχομένως και το Λουξεμβούργο, αν πρέπει και αυτοί να βάλουν το χέρι στην τσέπη, θα δυσκολευτούν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη, να υλοποιήσουν μάλλον τη δημοσιονομική εξυγίανση. Εμείς θεωρούσαμε ότι με την εκχώρηση του Λουξεμβουργέζικου τμήματος της Δέξια θα είχε ρυθμιστεί το πρόβλημα για το Λουξεμβούργο. Αλλά στις 26 ε, Σεπτεμβρίου μία μέρα πριν δηλαδή, είπατε ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι εγγυήσεις το 55 δις, προσωρινές εγγυήσεις. Εγώ δεν είμαι διευθυντή της Δέξια, έτσι. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τους υπεύθυνου της Δέξια και από τα κράτη, είτε που δανείζουν εγγυήσει ε, ή που ασχολούνται με τις εγγυήσει. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Τι κάνει η Κομισιόν. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο των κρατικών ισχύσεων, αναλύει την ε, πώληση της BIL στο Κατάρ κατά 90%. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό. 730 δις, έτσι. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Εμείς είπαμε ότι η ευθύνη μας είναι να λύσουμε το, το κομμάτι κρατικές ενισχύσεις. Και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Και είπα στον Υπουργό, του είπα, Λουκ, εγώ δεν σου βάζω κανένα πρόβλημα. Από πλευρά μου είναι οκ το πράγμα. Για τα υπόλοιπα δεν είμαι υπεύθυνο. Για τι εγγύησει τώρα. Οι εγγύησει. Μέχρι την υιοθέτηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης από τη μία του ομίλου Ντέξια και το, το τμήμα της διατεταγμένης διάλυσης ή εξυγίανση του, του τμήματο 16 υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου να δανείσουν κάποιες κρατικές εγγύησεις. Και εμείς έχουμε την ε, ευθύνη να πούμε το ok, αν μπορούν να δοθούν αυτές οι εγγύησεις. Δεν έχουμε ακόμα τελική απόφαση για την ε, αναδιάρθρωση και την διατεταγμένη διάλυση. Και μια και δεν έχουμε τελική απόφαση, δεν μπορώ να πω δεν σας επιτρέπουμε να δώσετε αυτές τις κρατικές ε, εγγύησεις. Δώσαμε προσωρινές άδειες για αυτές τις εγγύησεις. Δεν είναι κάτι που θα προτιμούσα εγώ. Θα προτιμούσα να είχαμε την τελική συμφωνία και το περιμέναμε, αλλά πρέπει να περιμένω εγώ. Πρέπει να περιμένω τις προτάσεις, πρέπει να περιμένω τα σχέδια. Πρέπει να περιμένω να ακούσω τις ε, θετικές και αρνητικές γνώμες για την αναδιάρθρωση παύλα διάλυση του ομίλου Ντέξια. Αυτές οι προσωρινές κρατικές εγγύησεις ε, που παρατείνονται μέχρι τον Ιανουάριο με βάση τη συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών, ακόμα και αν το Λουξεμβούργο δεν είναι πια μέτοχος του ομίλου δέξια, το Λουξεμβούργο συμμετέχει ως ένα ποσοστό 3-4%, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό. Το μεγαλύτερο τμήμα όμως ανήκει στο Βέλγιο, 60%, μετά είναι η Γαλλία και το πολύ πολύ μικρό αυτό τμήμα ανήκει στο Λουξεμβούργο. Δεν επιβάλλαμε εμείς αυτή την ε, συμφωνία, ούτε την ε, εγκρίναμε. Τα τρία κράτη συμφώνησαν. Οι τρεις κυβερνήσεις αποφάσισαν αυτή την κατανομή κάποια στιγμή. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν θέλω να χρεοκοπήσω ο φίλος μου, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Και δεν μπορώ να πω μια μέρα, τέρμα, δεν δίνουμε πλεονάτια για προσωρινές ε, κρατικές εγγύησεις, γιατί δεν είσαστε σε θέση να προβείτε στο τελικό σχέδιο της αναδιάρθρωσης διάλυσης. Απλώς θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να τραβήξει πολύ, γιατί ούτως ή υπάρχουν ζημιές και πρέπει να υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση αυτή τη τράπεζα αυτού του ομίλου. Ποιο θα πληρώσει, θα πρέπει οι φορολογούμενοι αυτών χωρών που είναι οι μέτοχοι του ομίλου Ντέξια να βάλουν τα λεφτά. Ελπίζω του επόμενου μήνες όμως να βρεθεί η λύση για αυτό το θέμα. Και για το θέμα της ε, στατιστικής μεταχείρισης από πλευράς Eurostat, όταν ήμουν πιο νέος ήμουν υπεύθυνο για αυτά τα θέματα. Τώρα ο Αλγύρντα Σεμέτας είναι επίτροπος για τελωνία, για σχέσεις με στατιστικές υπηρεσίες και με Eurostat. Αυτός είναι υπεύθυνος, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Eurostat. Ελίσσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Τρία ερωτήματα. Η πρώτη έχει να κάνει με τις πρακτικές που είναι όλο και πιο βίαιες μέσα σε αυτό το κρίμα, στο κλίμα κρίσης από τις αλυσίδες διανομής των τροφιμικών κυρίως προϊόντων. Δεν έχουν λειτουργία μόνο σε εθνικό επίπεδο, λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να συντρίβουν πλήρως τους μικρούς παραγωγούς εφαρμόζοντας πάρα πολύ σκληρούς όρους πληρωμής των προϊόντων, πιέζουν τις τιμές του παραγωγού και έχουν μια σαφή δεσπόζουσα θέση στις εθνικές αγορές. Θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν έχει την πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο σε σχέση με τα δίκτυα δανομής για να αντιμετωπιστεί αυτό το ερώτημα. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τις ε, περιφερειακού χαρακτήρα επιδοτήσεις. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία για τα θέματα αυτά. Ενώ σκεφτόμαστε λοιπόν για την μεσοπρόθεσμη δομή της Ευρώπης και έχουμε τις ε, εκθέσεις του Φαν Ρομπέι ή των τεσσάρων πρόεδρων, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να μπει μέσα στα σκαριά κάποιο είδος συνεργασίας των φορολογικών αρχών και των φορολογικών πολιτικών σε σχέση με τους συντελεστές που ακολουθεί κάθε χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άγριος ανταγωνισμός που ισοδυναμεί με δημοσιονομικό ντάμπινγκ και οδηγεί στο ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Και το τρίτο ερώτημα δεν αφορά την τέξια συγκεκριμένα, αλλά γενικά στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Προχωρούμε προς την κατεύθυνση μιας τραπεζικής ένωσης, η οποία θα περιλαμβάνει ένα επόπτη για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες που βρίσκονται σε φάση επανακεφαλαιοποίηση και ενδεχομένως και σε φάση επίλυσης. Επομένως, <clears throat> εδώ θέλουμε να έχουμε μία ενιαία εποπτεία, αλλά θα αφήσουμε τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης και ενδεχόμενης επίλυσης πάλι θα τα αφήσουμε στα χέρια των εθνικών αρχών επίλυσης. Και πάλι φυσικά θα χρησιμοποιήσουν χρήματα των φορολογούμενων για την ανακεφαλοποίηση αυτή ή την επίλυση και φυσικά κάθε χώρα έχει διαφορετική οικονομική δυνατότητα στην υποστήριξη αυτών των τραπεζών. Κάτω από ποιε προποθέσει λοιπόν ο μηχανισμό σταθεροποίηση, το ESM, θα μπορέσει να παρέμβει σε αυτέ τι περιπτώσει και τέλο η Κομισιόν θα δεχόταν να αναλάβει την, αρμοδιότητα επί, επίλυσης των τραπεζών γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ναι, θα απαντήσω στα ισπανικά βέβαια. Για τον τομέα της διανομής. Ναι. Δεν αρνούμε την πιθανότητα να υπάρχουν περιπτώσεις όπου να απαιτείται μια παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε βρεθεί ενώπιον μιας τέτοιας περίπτωσης. Ίσως η task force που έχουμε θέσει σε λειτουργία και η οποία βασίζεται στην εμπειρία, στην κτηθήσα εμπειρία και τις ε, περιπτώσεις που αντιμετωπίσαν οι εθνικές αρχές ε, ανταγωνισμού μέσα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού, ίσως θα μπορέσει να προκύψει μια νέα πρωτοβουλία. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάποια πρωτοβουλία σε, εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός αν υπάρχει κάποιο παράπλευρο πρόβλημα όπως παραδείγματος χάρη ήταν η συσκευασία ορισμένων τροφιμικών προϊόντων, ένα θέμα αρκετά περιθωριακό το οποίο αντιμετωπίσαμε. Αλλά για τις πρακτικές του τομέα αυτού μέχρι στιγμής βάσει των αναλύσεών μας και των ερευνών που είναι σε φάση εθνικό, εμείς δεν έχουμε λόγο παρέμβασης. Δεν το αποκλείω το δημοσιονομικό ντάμπινγκ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Οι συνθήκες όμως τι λένε και βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λένε ότι όπως μέσα στα σύνορα κάθε χώρας μπορεί να υπάρξει μία διαφορά, όπως μέσα ε, σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υπάρχει διαφοροποιημένη αντιμετώπιση με τη φορολογία και πάρα πολλές φορές έχουμε ε, αντιταχθεί σε εθνικές επιδοτήσεις για να μην υπάρχουν διακρίσεις στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν θεωρεί ότι οι διαφορές φορολογίας μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με το μηχανισμό αντιμετώπισης των κρατικών επιδοτήσεων. Μόνο νομοθετικά θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και δυστυχώς η νομοθεσία για τα φορολογικά θέματα υπόκειται στον κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβουλίο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Πάρα πολλές φορές όταν είναι φανερό ότι υπάρχουν στρεβλώσεις μέσα στην εσωτερική αγορά δεν μπορούμε να δράσουμε γιατί οι συνθήκες και η νομοθεσία δεν μας το επιτρέπουν. Και το να εξαλείψουμε αυτή την πολυπικιλία φορολογικών ρυθμίσεων, αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με μια απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να, γίνουν πάντα, να γίνονται πάντα αλλαγέ συνδικών για να λύνουμε τα προβλήματα, αλλά για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα θα έπρεπε να πω ότι χρειάζεται μια αλλαγή συνθήκων για το θέμα αυτό η οποία είναι κατεπίουσα. Και τέλος συμφωνώ ότι πράγματι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ανισομέρειες όταν προχωράει με μεγάλη ταχύτητα ο ενίος επόπτης για τις τράπεζες, ενώ συγχρόνως δεν έχουμε προχωρήσει παράλληλα με το σύστημα εγγυήσεως τραπεζικών καταθέσεων. Συμφωνώ, είναι σαφές ότι αν έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς προόδου στις τρεις, στους τρεις πυλώνες της ε, Τραπεζικής Ένωσης, θα έχουμε αρνητικές απόρριες, θα έχουμε στρεβλώσεις και ενδεχομένως θα δημιουργήσουμε και περισσότερα προβλήματα από ό,τι προσπαθούμε να επιλύσουμε με την ιδέα που εγώ την ενστερνίζομαι το να έχουμε μια τραπεζική ένωση. Για το να λάβει η Κομισιόν την εξουσία της επίλυσης, εγώ δεν έχω καμία άποψη για το θέμα αυτό. Όπως σας είπα, η Κομισιόν δρά σαν μια de facto αρχή επιλύσεως, χρησιμοποιώντας μέχρι τα όρια των δυνατοτήτων της όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχει για τον έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων. Υπάρχουν όμως σαφή όρια, όπως είδαμε για την τέξη. Αν ήμασταν μια αρχή επίλυσης, θα είχαμε <clears throat> επιφέρει εμείς μια ε, συντεταγμένη επίλυση και διάλυση του ομίλου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πράξουμε. Ο Βέμαρ. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Καλώ ήρθατε άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω να ρωτήσω σύντομα μερικά πράγματα. Διαβάσαμε στην εφημερίδα ΕΛΠΑΗ στι 5 Οκτωβρίου ότι η τράπεζα Σανταντέρ και η Κάσα είναι οι πιο μεγαλύτεροι επενδυτέ τραπεζικοί. εσεί που είσαστε για τον ανταγωνισμό, αν είναι οι κύριοι μέτοχοι, Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Έπειτα πριν από τέσσερις ε, μήνες Μεταξύ των διαφόρων προϋποθέσεων υπήρξε και άλλη για τη συμμετοχή στις ε, τράπεζες που σώζονται πριν ε, φτάσουν εκεί τα χρήματα από το κράτος. Στην περίπτωση της Μπάνκια τι ισχύει. Και εδώ έρχομαι και στην ερώτηση που έκανε και ο συνάδελφος Έπινγκ. Σας ρωτάω, έχει κανείς την εντύπωση ότι διάφορες μικρές ε, αποταμιευτικές τράπεζες της Ισπανίας αναγκάστηκαν σε εξυγένση και πουλήθηκαν ε, στη Μεγάλη Ισπανική Τράπεζα. Η δημιουργία της Μπάνκια ε, λοιπόν με τη συγχώνευση διαφόρων τέτοιων μικρών τραπεζών δημιούργησε μια μεγάλη τράπεζα του Big to Fail και αποφάσισε να την εθνικοποιήσει η κυβέρνηση και κάτι πιο επίκαιρο. Χτες έπαιξαν η Μπαρθελώνα με την Ρεάλ Μαδρίδ και εγώ παρευρέθηκα εκεί στο γήπεδο. Η Ρονάλντο και ο Κάκα πριν από μερικά χρόνια, ένας με 9 δισεκατομμύρια και άλλος με 60 δισεκατομμύρια ε, πουλήθηκαν ή υπάρχουν ε, αυτές οι συναλλαγές στην σε διάταξη ή τελικά τα χρήματα του φορολογούμενου χρηματοδοτούν μια θέμητη, έναν αθέμητο ανταγωνισμό στον αθλητικό τομέα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, λέει ο κύριος Σαλμούνια, μια που με ενδιαφέρει πιο πολύ καθότι ποδοσφαιρόφιλος. Θα ήθελα να δω η Bayer ε, Μούνικ πώς χρηματοδοτεί την αγορά του παίκτη της. Πριν έλεγα ότι δεν είμαι υποψήφιος για υπουργό στέγασης της Ολλανδίας, ούτε βέβαια και υποψήφιος είμαι για υπουργό οικονομικών της Ισπανίας ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, δεν ε, πρέπει εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές. Άλλοι υπουργοί, παλιότεροι, σημερινοί, οι ε, διοικητές τραπεζών πρέπει να απαντήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι το να συμμετέχουν κάποιες τράπεζες ε, στα μετοχικά κεφάλαια, αυτό είναι θέμα των ε, διοικητών και των αναλύσεων που κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, εκεί δεν υπάρχει τίποτα ούτε υπέρ ούτε κατά μια τέτοια δυνατότητες. Τώρα η πώληση ε, σε τράπεζες οι οποίες ε, βρίσκονται σε αναδιάρθρωση. Αυτό το οποίο διαπραγματευόμαστε και γι' αυτό είμαι εγώ υπεύθυνο είναι τα σχέδια αναδιάρθρωσης των δημοσιονομικών οντοτήτων ισπανικών που επειδή χρειάζονται κεφάλαιο και δεν μπορούν να έχουν από τις αγορές το κεφάλαιο αυτό, θα χρειαστούν μία ένεση δημοσίου χρήματος κεφαλαίων από το μηχανισμό που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή ένα δάνειο διευκόλυνσης το ΦΡΟΠ και το ΦΡΟΠ μπαίνει στο κεφάλαιο των οντοτήτων αυτών που δεν μπορούν να βρουν με άλλο τρόπο κεφάλαιο. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης που διαπραγματευόμαστε αποτελούν προϋπόθεση αναγκαία προκειμένου να πάρουν κρατικές ενισχύσεις, να πάρουν χρήματα από το κράτος μέσω του μνημονίου κατανόησης. Και σε αυτά τα προγράμματα αναδιάρθρωσης να ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ. Διαπραγματευόμαστε ήδη για την Μπάνκια, για την Καταλούνια ε, το Ποτεμιευτήριο, της ε, Γαλλικίας και της Βαλένθια. Είναι οι τέσσερις οντότητες που εθνικοποιούνται από το ΦΡΟΠ. Στην περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή του κλάδου πρέπει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. αν πρέπει να γίνουν επενδύσεις ή όχι, όταν να συμφωνήσουμε τα προγράμματα αναδιάρθρωσης, θα είναι εντελώς δημόσιες οι αποφάσεις και διάφανες. για τη δημιουργία της Μπάνκια αυτό που είπα και στον κύριο Έπινγκ. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Ήταν μια απόφαση που πήραν οι Ισπανικές αρχές τότε. Τώρα να προσθέσω και κάτι σε αυτά που είπα στον κύριο Έμπινγκ, να που μιλάω τώρα Ισπανικά. Υπήρξε τότε μια εγγραφή από το ΦΡΟΠ για τον πεθεά που τώρα έγινε κεφάλαιο ήταν μια γραφή που ήταν κάτω από κάποιο επίπεδο πάνω από το οποίο χρειαζόταν ειδική κοινοποίηση. Εγκρίθηκε από τις Ισπανικές αρχές. Άπαξ και εμείς είχαμε εγκρίνει το γενικό ε, σχέδιο, μια που ήταν κάτω από το 2% του ενεργητικού κτλ. Και τελικά τώρα, αυτό που τώρα διαπραγματευόμαστε με τις ισπανικές ε, αρχές, θα αναλυθεί και θα εγκριθεί, θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, τις επόμενες ε, εβδομάδες για τις μετατρέψιμες. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που εγώ το χάσα το πρέπει να ήταν καταπληκτικό. Η ομάδα μου εμένα δεν έπαιζε πάντως χθες. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα για το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που δωστάνε. Έχετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Ωραία. Τότε. Έληξε η συνεδρίαση. Και σας υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί συνεδριάζουμε στην 3 ε, σε Κάποια άλλη επιτροπή χρειαζόταν την αίθουσα αυτή και γι' αυτό αλλάζουμε αίθουσα αύριο το πρωί. Θα τα ξαναπούμε αύριο.